Καλημέρα σας κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχηθώ το καλώς ορίσατε στους κυρίους Χόγκερβορστ και Λίκανεν. Ο κύριος Χόγκερβορστ είναι επικεφαλής του Διεθνού Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων, οργανισμού ιδιωτικού δικαίου που ρυθμίζει και ευθυγραμμίζει τα IFRS. Είχε, έχει περάσει από διάφορες θέσεις στο, στην Ολλανδική κυβέρνηση και ήταν και υπουργό Οικονομικών. Και ο κύριος Λίκανεν, που είναι ο νέος πρόεδρος του Ιδρύματος IFRS από τον περισμένο Οκτώβριο. Τον κύριο Λίκανεν τον γνωρίζετε και ως διοικητή της Τράπεζας της Φιλανδίας και επίσης μέλος του Διεθνούς ε, Νομισματικού ε, Ταμείου, του Συμβουλίου δηλαδή, και του ε, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επίσης Υπουργός Οικονομικών της Φιλανδίας, πρώην Επίτροπος και δυστυχώς τον χάσαμε από Ευρωβουλευτή. Εδώ θα συζητήσουμε σήμερα τις δραστηριότητες του IASP και το IFRS Foundation Trustees και ως γνωρίζετε έχουμε ένα ε, μέγα αριθμό θεμάτων που μας απασχολούν, το IFRS 17 που είναι τα πρότυπα για τις ασφαλίσεις, επίσης ασφαλιστικά συμβόλαια και ε, στην πραγματικότητα μια πρώτη απογραφή του Financial Reporting του IFRS 9. Άρα είναι πλήρες το πρόγραμμά μας και να αρχίσουμε δίνοντας το λόγο στον κύριο Γόγκερβολστ. Α, είχα στι σημειώσει μου ότι πρόκειται να μιλήσει ο κύριο Γόγκερ Φώστα. Ευχαρίστω να μιλήσει ο κύριο Λίκανε. Κύριε Πρόεδρε, πολύ χαίρομαι που επανέρχομαι στην Επιτροπή σα, όπου πριν από Λίγα χρόνια μιλούσαμε για τις αναδιαθρώσεις τραπεζών, ήδη από το 2002 και 2003, γιατί ήμουν μέλος της Επιτροπής που υποστήριξε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πρότυπα IFRS. Ταυτόχρονα υπήρχαν και δύο θέματα καινούρια. Τα αφενός ήταν το διαδίκτυο, το δεύτερο ήταν το IFRS, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με παρόμοιες προκλήσεις και αυτά είχαν εξελιχθεί στον ιδιωτικό τομέα με ε, πολύ καινοτόμες ε, λύσεις για τις αγορές, για την ψηφιακή πληροφορία και για την ροή των ε, οικονομικών πληροφοριών. Είχαν υπήρξε, υπάρξει τότε κάποιες ιδέες για τη δημιουργία ευρωπαϊκού διαδικτύου. Είχαμε πει τότε ότι η Ευρώπη τελικώς θα φτιάξει τη δική της εκδοχή των IFRS. Τελικώς υποστηρίξαμε τα IFRS με ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τότε δηλαδή ξαναλέω το 2002. Οι τραστείς, οι καταπιστευματοδόχοι είναι υπεύθυνοι για τη στρατηγική, για τους διορισμούς και για την διαχείριση του οργανισμού. Στην αρχική μας δήλωση λέμε ότι η διαφάνεια επιτρέπει στους επενδυτές να λάβουν αποφάσεις με, έχοντας την ε, διάθεσή τους αναγκαίες πληροφορίες. Η λογοδοσία κλείνει το κενό ανάμεσα στις ε, επενδυτικές εταιρείες και στην κοινωνία και αυτό είναι σημαντικό για τη διαχείριση. Τρίτο, αυξάνει την οικονομική αποδοτικότητα και βοηθεί τους επενδυτές να αναζητήσουν ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο και τέλος όταν εφαρμοστούν σωστά τα πρότυπα μειώνουν το κόστος του κεφαλαίου που σημαίνει επίσης ότι διευκολύνουν την, αύξηση, την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια και έχω κι άλλη μία. Ε, ε, μάλλον προχωρούμε άλλη μία. Δύο σχόλια τα οποία έχουν ε, έντονο χαρακτήρα και τα θυμούμε καλά σε όλη αυτή την υπόθεση των IFRS. Το 2002 είχαμε ε, επισκέπτη από τις Ηνωμένε Πολιτείε τον Πολ Βόκερ, πρώην πρόεδρο της Fed, ο οποίος ήρθε και έκανε μια ομιλία και θα θυμίσω τι είπε. Είπε τότε ότι εάν πρόκειται να, να λειτουργήσουν τα πρότυπα, οφείλουμε να σεβαστούμε τρία στοιχεία. Επαρκή διαβούλευση, να ακολουθούνται οι καθιερωμένες διαδικασίε λήψη αποφάσεων και τέλο να είναι γερά θεμελιωμένε. Αυτέ οι τρει αρχέ εξακολουθούν να ισχύουν και βεβαίω εδώ στην Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο επίση παίζει ένα ρόλο στην ε, καθιέρωση αυτών των διαδικασιών. Δεύτερο ομιλητή που άκουσα τον Νοέμβριο όταν για πρώτη φορά συμμετείχα ε, στην πρώτη συνεδρίαση ε, πιστευματοδόχος τραστή δηλαδή από την Νότια Αφρική ο σοφός Νουκούλου πρώτος ε, λογιστής στη χώρα του και είπε τότε το σύστημα IFRS είναι πολύ σημαντικό για την Αφρική διότι είναι το κρίσιμο πλαίσιο για την διαφάνεια των αλλοδαπών επενδύσεων που θα επιτρέψει στις κυβερνήσεις η διαφάνεια αυτή να αντιμετωπίσουν την διαφθορά. Αυτό είναι η αρχή και το τέλος αυτής της ιστορίας και είναι σημαντικά τα σχόλια αυτά για να κατανοήσει κανείς την πορεία αυτή. Έχω μια διαφάνεια ακόμη και το τελευταίο μου σχόλιο είναι για τα στρατηγικά θέματα διότι αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα των τραστής. Μόλις ε, συναντηθήκαμε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας τον Γενάρη και ξεκινήσαμε με ένα στρατηγικό προβληματισμό με τρία επίκεντρα ε, θέματα. Αφενός την απειλή της αποπαγκοσμιοποίησης, δεύτερο πώς να παραμείνουμε ε, σημαντικοί, τρίτο τι θα σημάνει η εξέλιξη τεχνολογίας για μας. Πολύ λίγα σχόλια για καθένα από τα τρία αυτά. Όλοι είδαμε ποιες είναι οι εξελίξεις ε, σε αυτή την τάση από παγκοσμιοποίησης που τη βλέπουμε σε, πολλές, ε, σε τομείς. Εμπόριο, για παράδειγμα. Έχει λιγότερο επηρεαστεί ο χώρος των προτύπων από άλλους τομείς. Χρειάζεται όμως να βασιστούμε στις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Διότι η τεχνολογία δεν πρόκειται να φύγει, ε, η ελεύθερη διακίνηση ε, κεφαλαϊκών αγαθών δεν πρόκειται επίση να σταματήσει, έστω και αν εγερθούν κάποια εμπόδια στο διάβα του. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πιο σημαντικό για μα να διασφαλίσουμε τον ρόλο των προτύπων με υψηλό επίπεδο διαφάνεια, λογοδοσία και αποδοτικότητα. Και αυτό είναι το καθήκον μα. Το δεύτερο είναι για τη λεγόμενη relevance, δηλαδή να παίζουμε σημαντικό ρόλο. Τα IFRS παίζουν σημαντικό ρόλο στο finance reporting γνωρίζουμε ότι οι επενδυτές επιθυμούν να γνωρίζουν περισσότερα σήμερα. Εάν συναντηθείτε με επενδυτέ, λένε θέλουμε να ξέρουμε βέβαια τα νούμερα σχετικά με την απόδοση των κεφαλαίων μα, θέλουμε να ξέρουμε όμω και άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Και έχουν βέβαια τα πράγματα αυτά και μακροπρόθεσμη ε, ε, απόδοση. Βιωσιμότητα, επίση κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε, μακροπρόθεσμα, πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. και πώς θα προσαρμοστούν στο ε, περιβάλλον ESG. Και ο ISP εργάζεται στον τομέα αυτό, θα τα πούμε και σε λίγο αυτά. Τρίτο είναι η τεχνολογία που ε, σας είπα ήδη από το 2000 μας απασχολεί. Βεβαίως και κινείται προς τα εμπρός. Αλλάζει τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούμε, με τους οποίους οργανώνουμε τις δραστηριότητές μας. Και για παράδειγμα, στον χώρο των προτύπων, όλο και περισσότεροι ρυθμιστές ανά τον κόσμο τώρα πλέον προχωρούν σε ηλεκτρονικό filing και σε άλλες ηλεκτρονικές δραστηριότητες. Και το σύστημα IFRS μπορεί να προσφέρει υψηλή ποιότητα ηλεκτρονική ταξινόμηση, ταξόνομη. Άλλο θέμα είναι βέβαια ποιος θα είναι ο ρόλος όλων αυτών των τεράστιων ε, όγκων δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Ποιο θα είναι ο ρόλο, μάλλον πόσο θα χρειάζονται οι επενδυτέ, με αυτή τη μάζα δεδομένων αν θα χρειαστούν κάποια ταξινόμηση και είμαι βέβαιος ότι ο σημαντικός ρόλος των IFRS θα παραμείνει, των προτύπων δηλαδή. Και βεβαίως και χρειάζεται και περισσότερες πληροφορίες και χρειάζεται να το παρακολουθούμε. Όσον αφορά το Ίδρυμα. Βεβαίως η ψηφιοποίηση είναι μια πραγματικότητα και είναι σημαντικό και το IFRS Foundation να περάσει στην ψηφιοποίηση. Έχουμε ξεκινήσει ήδη ένα μείζον πρόγραμμα ψηφιοποίησης των εσωτερικών συστημάτων μας και εξετάζουμε την ψηφιακή εμπειρία την οποία μπορούμε να προσφέρουμε και στους πελάτες μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και είμαι στη θέση σας για συνεργασία και στο μέλλον. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Λίκανεν. Θα δώσω τώρα το μικρόφωνο στον κύριο Βόρστ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή και ο χρόνος πιέζει, γι' αυτό θα σας μιλήσω κάπως σύντομα όσον αφορά τον Εργασμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και μετά φυσικά είμαι και στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Λοιπόν, ας πάμε στην διαφάνεια 7, η οποία τι δείχνει, δείχνει ότι είναι μια προτεραιότητα για την ε, κοινότητα, την ε, διεθνή, και ότι υπάρχει μεγάλη πίεση πάνω στα business models. Τώρα εννοείται ότι σε αυτό το IFRS 17 ε, πολλές φορές μειώνονται τα επίπεδα όπως στην Κορέα για παράδειγμα ακριβώ γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι η διαφάνεια βέβαια θα προσφέρει περισσότερη σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η επόμενη διαφάνεια 8 δείχνει τι κάνουμε εμείς στο στάδιο υλοποίηση. Πάνω από 20 θέματα έχουν εντοπιστεί στο στάδιο αυτό της υλοποίηση. Και είπαμε ότι θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας αλλαγές, αρκεί βέβαια αλλαγές να μην διακόπτει και να μην δρά αρνητικά στη διαδικασία αυτή υλοποίησης. Όπως γνωρίζετε ίσως από τα 27 θέματα υπάρχουν 6 κυρίως που έχουν εντοπιστεί από το ΙΦΡΕΓ αλλά και από άλλα σημεία του κόσμου και τους τελευταίους μήνες το Συμβούλιο αποφάσισε 6 αλλαγές στις προδιαγραφές από τις οποίες πέντε διακόπτεται το μικρόφωνο του μιλητή. Θα έπρεπε να είναι σαφές στο κλάδο ποια πορεία θα ακολουθήσουμε. Μερικές φορές μειώνονται θέσεις, υπάρχει μετάβαση, υπάρχουν τα δάνεια τα οποία αναμειγνύονται με ασφαλιστικά προϊόντα, όμως εμείς ανταλαμβανόμαστε ότι έτσι κι αλλιώς το χρονοδιάγραμμα ήταν πολύ σφιχτό και σκεφτήκαμε ότι μια τέτοια αλλαγή καλύτερα αντί για το 2021 να γίνει το 2022. Και βέβαια παρόλο που πολλοί ασφαλιστές θέλανε περισσότερο χρόνο, θα σας το πούν, από την άλλη είναι ευτυχή που η παράταση δεν είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί υπάρχει ένα ρυθμό που ακολουθούμε και όσο περισσότερο κρατήσει υλοποίηση, τόσο περισσότερο θα κοστίσει κιόλα. Τέλος, να σας πω και δύο λόγια για το ρόλο του SB στην ε, χρηματοπιστωτική αναφορά. Και ξέρω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η αναχώρα συστάσεις. Σας είπα νωρίτερα ποιο είναι το έργο μας προκειμένου να ανανεώνουμε τα σχόλια, να τα ενημερώνουμε και βοηθάμε τις επιχειρήσεις για το πώς θα ετοιμάζουν τις ετήσιες εκθέσεις τους. Σε αυτές μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα που είναι κατάλληλα χρηματοπιστωτικά, αλλά από την άλλη μεριά δεν ανήκουν στις χρηματοπιστωτικές αναφορές, όπως είναι τα business models και πληροφορίες για το μέλλον, προβλέψεις δηλαδή. Αυτό που είναι επίση σαφέ είναι ότι υπάρχουν όλο και περισσότερο θέματα βιωσιμότητα, γιατί υπάρχει η κλιματική αλλαγή. Τι οικονομικέ συνέπειε θα έχει στι επιχειρήσει αν δουλεύετε στον ενεργειακό τομέα, στην εξόριξη, η κλιματική αλλαγή, τα περιβαλλοντικά μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Οπότε τα διαχειριστικά σχόλια θα ήταν το κατάλληλο σημείο για να γράψετε για αυτά ως επιχείρηση. Βοηθούμε λοιπόν ακριβώς να υπάρξει αυτή η ενημέρωση στα σχόλια ώστε να είναι πιο κατάλληλα επί τόσον αφορά τις στρατηγικές. Και αυτές μπορεί να επηρεάσουν ε, την ε, μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα και είναι και αυτό κάτι που μπορεί να διατυπώσει κανείς στην ετήσια έκθεση. Τέλος θα σας μιλήσω για το θέμα των αναχώρας συστάσεων. Στην προηγούμενη συνάντησή μας σας είχα πει ότι θα συνομιλούσα για αυτό το θέμα με τις υποπτικές αρχές για να δούμε κατά πόσο είναι κάτι που πρέπει όχι να γίνει. Συζητήσαμε λοιπόν αρκετές φορές με το ε, Εποπτικό Συμβούλιο για να δούμε τι είναι καλύτερο και η δικιά μας η θέση ήταν, όπως το έχω ξαναπεί και εδώ, ότι δεν πιστεύουμε ότι το IFRS συνδέεται άμεσα και πάει παράλληλα και αναλογικά με το με τις αναχώρες συστάσεις. Είναι πληροφορίες που είναι, πιστεύουμε, εκτός πεδίου χρηματοπιστωτικών αναφορών. Έπειτα, ο ορισμός του εισοδήματος είναι διαφορετικός. Οπότε, εμείς είπαμε στο Εποπτικό Συμβούλιο ότι η νέα δήλωση των διαχειριστών όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές αναφορές, οι στρατηγικές θα μπορούσαν απλώς ίσως να κάνουν μια σύνδεση ανάμεσα στις αναχώρα συστάσεις. Ακόμα και αν και σε άλλες περιπτώσεις τις προδιαγραφές τις σχετικές δεν τις κάνουμε εμείς. Φυσικά είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και τον ΩΣΑ εφόσον χρειάζεται από εμά κάποια βοήθεια για την διατύπωση. Τώρα νομίζω ότι θα ήταν δίκιο επίσης να πούμε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο να σας πω, είχαμε πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων, αλλά οι απόψεις τους διαφέρουν, να ξέρετε, μεταξύ τους. Δεν καταλήγουν σε επίσημη θέση. Πιστεύω όμως ότι συζητήσαμε καλά και ότι κατανόησαν τα δικά μας επιχειρήματα. Και στο τέλος μας ικανοποιεί η θέση την οποία υιοθετήσαμε που είναι να μην ασχοληθούμε με τις ε, χώρα συστάσεις, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα κάποιου σχολείου εφόσον υπάρξουν κάποιες επικίνδυνες στρατηγικές. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου, Πρόεδρε, και από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας. Και τώρα οι συνάδελφοι έχουν τον κύριος Στόλογεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χούκερβόστ, τον πρώην πρόεδρο του του του Ιδρύματος ΕΦΕΡΕΣ και τον, τον κύριο Πράντα και, τον, ε, και για τη συνεργασία μας κατά τη διάρκεια όλης αυτής της θητείας. καταφέραμε πολλά σημαντικά πράγματα για το ΕΦΡΕΣ, όπως ε, τις ε, συμβάσεις, τα τραπεζικά, το leasing. Έγινε πολύ καλή δουλειά από όλους και ελπίζω ότι στην επόμενη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα αποφασίσει αυτόν τον μόνιμο διάλογο και την συνεργασία μας για τα θέματα ARS, αεφερές να τη διατηρήσει. Πέραν αυτού, θέλω να θέσω κάποια θέματα ή ερωτήσεις τέλο πάντων. Το πρώτο είναι τα συμβόλαια τα ασφαλιστικά. Όπως ξέρετε, ήδη κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, ιδίως αντασφαλιστικές, μας έχουν αποστείλει επιστολές και απογοητεύτηκαν με το ψήφισμα που μόλις αναφέρθηκε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι είδους διαδικασία σκοπεύετε να ακολουθήσετε για να προσπαθήσετε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα που αναφέρουν οι εταιρείε, οι αντασφαλιστικέ, οι λεγόμενε MTL. Ε, το δεύτερο θέμα είναι αυτό που αναφέρατε για τη διαφορά μεταξύ της, των προτύπων υποβολής εκθέσεων για θέματα χρηματοοικονομικά και άλλα που επίσης βρίσκονται στον κατάλογο προτεραιότητων του Ευρωκοινοβουλίου, για τις εταιρείε ας πούμε, και για την κοινωνική διακυβέρνηση. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να μπερδέψουμε την υποβολή εκθέσεων για τα θέματα τα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά με άλλα, αλλά ήθελα και τις δικές σας τις απόψεις. Ήθελα λοιπόν να καταλάβω την άποψή σας για την υποβολή εκθέσεων και το θέμα της κοινωνικής διακυβέρνησης μας και μετά για τις εταιρείε τεχνολογικού περιεχομένου, τεχνολογικές εταιρείε τι προβλέπετε εσείς να κάνετε, ιδίως για τα άειλα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ε, ισολογισμό των ε, εταιριών αυτών. Έχετε κάτι στον κατάλογο των προτεραιοτήτων σας. Και σας ευχαριστώ και πολύ για όλη σας τη δουλειά αυτά τα χρόνια. Κύριε Στόλογιαν, πολύ ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Και για μα ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν πάντοτε απλέ οι συζητήσει μας, όμως υπήρχε άμεση και ανοιχτό μια επικοινωνία και πετύχαμε πολλά, όντω. Η μόνιμη ομάδα εργασίας ε, για το ΑΕΣ ήταν πολύ επικοδομητική ως δουλειά. Απόφαση του Κοινοβουλίου ήταν αυτό και ελπίζω όντως να συνεχιστεί και στο μέλλον για τα συμβόλαια ασφαλίσεων. Δεν γνώριζα το πρόβλημα των αντασφαλιστικών. Μάλλον έχει να κάνει με τα αξιόγραφα. Θα φροντίσω όμως τις σχετικές πληροφορίες να τις ε, επισημάνω στους συναδέλφους μου. για τις εξωοικονομικές ε, ε, πληροφορίες και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ε, η προείπα ότι δεν είμαστε έτοιμοι να καθορίσουμε πρότυπα για θέματα λόγου χάρη βιωσιμότητας. Χρειάζεται διαφορετική και τεχνική γνώση εδώ και είναι πολλές οι ενώσεις και οι οργανισμοί που ήδη κάνουν τέτοια δουλειά. Δεν χρειάζεται να πάμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Δεν θα εξυπηρετήσει σε κάτι. Ωστόσο, θέματα όπως τα περιβαλλοντικά, όπως είπα και στην εισήγησή μου, θα αποκτήσουν ιδιαίτερη οικονομική βαρύτητα και στο μέλλον σε σχέση με την βιωσιμότητα μιας εταιρεία, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί επαρκώς στις οικονομικές ε, εκθέσεις, στην οικονομική καταγραφή στοιχείων να απεικονιστεί αμέσως αλλά θα χρειαστεί λαμβάνεται υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν την καθοδήγησή μα την ε, ε, έχουμε προσαρμόσει ώστε να υπάρξει κάποιο είδου συνδυασμό τη καταγραφή τη βιωσιμότητα με την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων. Για το μέλλον μια εταιρεία οι επενδυτέ πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει και με τη βιωσιμότητα σε μια τύση έκθεση, λίγο πολύ. Δεν μπορούμε λοιπόν εμεί να δημιουργήσουμε τα πρότυπα. Ε, αλλά αν, α πούμε, μια εταιρεία κινδυνεύει από τι απειλέ των κλιματικών αλλαγών, πρέπει να είναι γνωστό είναι δουλειά τη ομάδα κρούση, ε, τη ομάδα δράση, μάλλον, συγγνώμη, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σχετικό σχόλιο στι δηλώσει της τώρα. Τα σχόλια του management τη διευθυντική ομάδα είναι το καλύτερο σημείο για να περιγραφούν τα άλλα περιουσιακά στοιχεία μια εταιρεία. Διότι στου ολογισμού Πολλέ φορέ γράφονται όλα τα στοιχεία για το μετρητό που είναι πολύ, αλλά αυτό που δεν εξηγούν είναι η τεχνολογία και η τεχνογνωσία και πώς αυτό αποτιμάται. Δεν είναι εύκολο να καταγραφεί τις οικονομικές δηλώσεις. Είναι πολύ σχετικές, αφηρημένες και θεωρητικές πληροφορίες. Είναι δύσκολο κανείς να τις καταγράψει πρακτικά και σε τι βαθμό φτάνουν. Δεν νομίζω λοιπόν οι εταιρείε να αρχίσουν να τα γράφουν αυτά στι οικονομικέ δηλώσει, όμω νομίζω τα σχόλια του management στι αιτήσει εκθέσεις θα μπορούσαν να εξηγούν ποια είναι η σχετική αξία των ε, τεχνολογικών ε, προόδων ή των τεχνολογικών κατακτήσεων μιας εταιρείας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Στόλογεν και τα άλλα μέλη της μόνιμης ομάδας εργασίας για, τα, για το IFRS. νομίζω είναι μια ομάδα που είναι πολύ χρήσιμη ε, και θα ήταν καλό να συνεχίσει να υπάρχει και στην επόμενη θητεία. Είναι καλό να έχει το Κοινοβούλιο μια ομάδα που να ασχολείται ειδικά με αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτή τη δυνατότητα ανταλλαγή πληροφοριών και διαλόγου. Περβάνη μπερές. Ευχαριστώ πολύ από τους σοσιαλιστές. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την ε, μόνιμη ομάδα εργασίας και για, το, για τη δουλειά του κυρίου Στόλογεν σε αυτήν την ομάδα. Χαίρομαι ιδιαίτερος που ξαναβλέπω τον κύριο Λίκανεν στη νέα του θέση, κρίσιμη σημασία. Και εδώ διάλογος με το κοινοβούλιο, του οποίο γνωρίζει όλους τους ε, δεδάλους, είναι τους λαβυρίνθους μάλλον, είναι πολύ σημαντικός. Ε, εδώ, για τις αντασφαλιστικές πάλι, θα, θα ζητήσω και εγώ να το κοιτάξετε πολύ προσεκτικά, γιατί για τις ασφάλειες έχουμε αυτό το πρόβλημα των αντασφαλίσεων. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Λυπούμε που κάνατε αυτή την για την, ε, ανακοίνωση για την αναχώρα υποβολή εκθέσεων. Υπάρχει εδώ κάποια αντίθεση δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο είδου συμφωνία με τον ΩΣΑ και πώ να διοργανωθούμε, αλλά εμεί, η δική μα πολιτική πεποίθηση, και είμαστε εδώ για να περάσουν και πολιτικά μηνύματα βεβαίω, είναι το θέμα είναι ότι, η υπόθεση του CBCR, ε, αν μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, θα είναι πρόβλημα. Είναι απαραίτητο για να υπάρχει η κατάλληλη φορολογική διακυβέρνηση και τη χρειαζόμαστε και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό. Είναι θεματάκι λοιπόν αυτό για μας. Το βασικό σημείο το οποίο θέλω όμως να σχολιάσω είναι η έκβαση της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου των εμπειρογνωμόνων και το τι είναι αναγκαίο στην Ευρώπη για να ληφθούν υπόψη τα μη οικονομικά κριτήρια στην καταγραφή των στοιχείων των επιχειρήσεων. Πώς μπορούν όλα αυτά να διαρθωθούν διότι λέτε ότι δεν είναι τίποτα καθοριστικό για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά πάρτε την ε, έννοια των ασφαλιών. Οι ασφαλιστικές είναι πλέον εκτεθειμένες. Ε, σκεφτείτε τι γίνεται με ένα stranded asset ή με το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι μέρος της βασικής δουλειάς μιας τέτοιας εταιρείας δεν μπορούμε να αναβάλουμε πάπυρον ε, την συμπερίληψη όλων αυτών και στην ε, λογική που ακολουθούμε και στην καταγραφή των στοιχείων μιας εταιρεία. Ιδίω εάν δούμε τα συμπεράσματα του, της ομάδας ψηλού ε, καταλήγουμε ότι και για το θέμα αυτό, εάν η Ευρώπη προχωρήσει πιο γοργά από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα λόγω χάρη, επιβάλλοντας, ξέρω εγώ, την καταγραφή τέτοιων στοιχείων, ιδίω και με το αρχιτεκτόνιμα το φορολογικό που θα φτιάξουμε, τότε ίσως ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε καρβινίν. Το ανάποδο δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει υπερβολικά. Βεβαίω, ε, θα μου πείτε υπάρχουν τα ανάλογα διεθνή πρότυπα και μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά εάν οι υπόλοιποι δεν προχωρήσουν αρκετά γρήγορα για να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο φορολογικό αρχιτεκτόνα που να λαμβάνει υπόψη τι ανάγκε και των χρηματαγορών και των ε, εταιριών για να δούμε τι θα κάνουμε τα stranded assets, ε, πρέπει κάποτε να κουνηθούμε. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιμένει. Αν όλοι δεν θέλουν να πάνε με τον ίδιο ρυθμό, θα πρέπει κάποιοι να μπορέσουν να πάνε στην πρωτοπορία εφόσον το θέλουν. Και να κάνουν και το κάρβινγκ που του χρειάζεται. Um, Πρώτα απ' όλα για την αναχώρα υποβολή εκθέσεων. πραγματικά το ανέλησα πολύ και στο Διευθυντικό Συμβούλιο, σας το είπα αυτό. Και, ε, και πραγματικά ανέπτυξα, ασχολήθηκα πολύ με το τι κάνει ο, ο και το μελέτησα και με εντυπωσίασε το πώς προχωρούν, ε, πόσο η συμφωνία έχει προδεύσει και πόσο ε, υπάρχει διεθνή συνένεση. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ευκαιρία. Διότι και στον ΩΣΑ Φαίνεται ότι η αναχώρα υποβολή εκθέσεων και καταγραφή στοιχείων αναχώρα απομονωμένα μπορεί να είναι πολύ παραπλανητική. Πρέπει να συνδυαστούν τα στοιχεία, να υπάρχει καταγραφή των συγκυριών και συνδυασμένε πληροφορίε. Δεν υπάρχει περίπτωση στο εγγύ μέλλον αυτό να γίνει δημόσιο, αποκλείεται. Είναι μια πορεία που υπόσχεται πολλά αυτή του ΩΣΑ για την ώρα και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι η δική μου η σύσταση, η δική μου προτροπή. Δεν θέλω να απεκδηθώ των ευθυνών, αλλά νομίζω ότι για την ώρα έχουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Για τη βιωσιμότητα και την καταγραφή των σχετικών στοιχείων. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται κανένα καρδί για να γίνει. Δεν είναι απευθεία δική μα ευθύνη. Ακόμη και με τα δικά μα τα πρότυπα και τι προδιαγραφέ, ακόμη και αν θελήσουμε κάτι, μπορούμε να προβλέψουμε την ανάλυτη όλη νομοθεσία για να καταστεί εφικτό αλλά ως προς την βιωσιμότητα στην Ευρώπη ε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε σίγουρα, αλλά ήδη κάνουμε κάποια πράγματα. Θυμηθείτε, τη συζήτηση την κάναμε και με την ε, συζήτηση για το FRS 90. Ξέραμε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που έχουν ακριβώς να κάνουν με την βιώσιμη ανάπτυξη. Και εδώ Αυτό που είχαμε δει πριν την υιοθέτηση του 90 ήταν ότι θα υπάρχει ε, η επίπτωση για το κάρβιν. Τώρα η μελέτη που, εκδόθηκε αποδεικνύει αυτό που λέγαμε. Δεν είναι τελείως άσχετα με την εφαρμογή του έφερε. Ναι, αλλά εδώ μιλάτε για δημοτικονομική καταγραφή στοιχείων και συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν. Εκεί σίγουρα θα χρειαστεί κάτι. Αλλά αυτό που είπατε για τι ασφάλειε είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι και δική μου πεποίθηση ότι οι ασφαλιστικέ είναι πάρα πολύ εκτεθειμένε στι ε, κλιματικέ αλλαγέ και είναι απειλή τώρα. Όμως η ουσία των τύπων που έχουμε δημιουργήσει είναι ότι ε, κοιτάνε σε πολύ μακρινό μελλοντικό ορίζοντα για να μπορούν να λάβουν υπόψη και απώλειες μελλοντικέ και εξελίξεις μελλοντικέ, όπως αυτές που θα προκαλέσουν οι κλιματικές αλλαγές. Νομίζω λοιπόν τα ε, πρότυπα μας όπως τα έχουμε αναπτύξει επιβάλλουν στις ασφαλιστικές να τα λάβουν αυτά υπόψη λαμβάνουν υπόψη ότι θα πρέπει να τα πληρώσουν, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη που θα πρέπει να επενδύσουν για να μπορέσουν να καλύψουν τα περιουσιακά τους. Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Δεν είναι μέρος του προτύπου μας, αλλά εάν υπάρχει κάποια επικάλυψη σε σχέση με την καταγραφή στοιχείων βιωσιμότητα, που δεν θέλουμε να την κάνουμε γιατί έχει πολλέ διαφορετικέ προεκτάσει και δεν μας, ε, ε μπορεί να μα ε, επιληθεί από εμά τώρα. Ε, εκεί που τα στοιχεία βιωσιμότητα μπορεί να γίνουν σημαντικά για την οικονομική διάσταση μια εταιρεία, την ευρύτερη οικονομική καταγραφή στοιχείων, εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Και σίγουρα μπορεί να υπάρχουν οικονομικέ επιπτώσει. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω από το ECR κανέναν, ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ πολύ. Μια που έχουμε και διερμηνία, την ερώτησή μου θα την υποβάλω στα γερμανικά. Ο κύριος Λίκανεν αρχικά μας είπε ότι 87% παγκοσμίω χρησιμοποιούν το IFRS. Το 2004 ο τότε γενικό διευθυντή του IFRS μου είχε πει ότι είναι ζήτημα λίγων μηνών και μέσα σε λίγου μήνε θα συμμετείχαν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα χρησιμοποιήσουν και αυτέ δηλαδή το IFRS. Ωστόσο, έχουν περάσει 15 χρόνια και οι Ηνωμένε Πολιτείε ακόμα δεν συμμετέχουν, ούτε η Κίνα. Και γι' αυτό η ερώτησή μου. Εάν οι δύο σημαντικότερε οικονομίε του κόσμου, δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε και Κίνα. Δεν χρησιμοποιούν το πρότυπο IFRS. E IFRS. Μήπως είναι ψευδέστηση να πιστεύουμε ότι όπου να είναι θα έχουμε ενιαία πρότυπα. Δεύτερο. Το ερώτημα, το μέγα ερώτημα είναι τι κάνουμε με τις λεγόμενες ψηφιακές επιχειρήσεις, ιδίως στη Silicon Valley που έχουν και παγκόσμιες ε, επιχειρηματικές δραστηριότητες και δεν είμαστε βέβαιοι επειδή είναι και προερχόμενες από τις Ηνωμένε Πολιτείε, επομένως στη χώρα τους δεν χρησιμοποιούν τα πρότυπα IFRS, θα δημοσιεύσουν τα νούμερά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε τελικώς να τις φορολογήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές. Γι' αυτό και ρωτώ τι μπορούμε να κάνουμε. Αρκούν οι δυνατότητες που προσφέρει το πρότυπο IFRS ώστε να μπορέσουμε να απεικονίσουμε τις αποδόσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φορολογηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέπτεται να εισαγάγει ψηφιακό φόρο. Αυτό όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φορολόγηση του κύκλου εργασιών. Στο μεταξύ υπάρχει και ένας αριθμός πολιτικών σχηματισμών που λένε ότι η απόδοση μιας οικονομίας δεν μπορεί ε, να απεικονίζεται μονάχα στο ακαθάριστο ε, εθνικό προϊόν. Υπάρχουν και άλλοι ποιοτικοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εάν είναι σωστέ οι σκέψει αυτέ, τίθεται το ερώτημα εάν αυτό οφείλει να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των επιχειρήσεων. Και υπάρχουν σχετικέ σκέψει στα πλαίσια του IFRS, δηλαδή σχετικά με διεύρυνση των κριτηρίων, ώστε να μετρηθεί πέραν από την top και bottom line ποσοτική ε, απόδοση, να λεβεληθούν και οι άλλοι παράγοντες. Και τελευταία ερώτηση, τα λεγόμενα εικονικά νομίσματα όπως bitcoin κλπ. Ποιες δυνατότητες έχει το πρότυπο IFRS να καταγράφει καταλήλως και να απεικονίζει στους λογαριασμούς τις δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ ε, έχω ασχοληθεί με τα εικονικά νομίσματα πρόσφατα. Τώρα για την Αμερική, αλλά θα τα απαντήσω ο Χόκερφορστ. Με Αμερική και, ε, και Κίνα. Ήδη είχαμε αρχίσει με τον Πολ Γόκερ, όπως είπαμε τότε, το 2002. Ήταν μια αρχική φάση της εξέλιξης και ήμασταν τότε πράγματι πολύ αισιόδοξοι, υπερβολικά αισιόδοξοι. Δυστυχώς δεν επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις αυτές. Ωστόσο υπάρχουν δύο θετικά σημεία Αφενός, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τα πρότυπα IFRS και δεύτερο, μίλησα πριν για την ταξινόμηση η οποία ε, χρησιμοποιεί το IFRS, ε, το ISB εδώ στην Ευρώπη. Υπάρχουν δηλαδή κάποια κοινά στοιχεία. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη εικόνα αλλά α δούμε και αυτή την θετική πλευρά, έτσι κι αλλιώ. Η Κίνα τώρα. Έχω συναντηθεί με τους Κινέζους ομολόγους για πολλά χρόνια. Και βλέπω δέσμευση τώρα της Κίνας, ίσως εντονότερη από ό,τι στο παρελθόν. Όταν συγκρίνω δηλαδή ισολογισμούς εταιριών, αυτών δηλαδή, όπως για παράδειγμα στο χρηματιστήριο του, του Hong Kong που χρησιμοποιούν δηλαδή το κινέζικο σύστημα και αυτό που χρησιμοποιούν το FRS. Είναι πολύ συγκρίσιμη η ισολογισμή αυτή. Στο κάτω τη γραφής, όσο προχωρεί η παγκοσμιοποίηση, θα θέλουν και αυτοί να δείξουν τι έχουν επιτύχει. Ίσως λοιπόν εδώ μπορούμε να δούμε περαιτέρω πρόοδο. Όμως για τα εικονικά νομίσματα καλύτερα να απαντήσει ο Γόγκερφορστ να συμπληρώσω κάτι για την Κίνα πρώτα. Οι επιχειρήσεις εκείνες που κάνουν dual reporting στο Hong Kong, 200 από αυτέ έχουν ταυτόσιμες ταυτόσιμους ισολογισμούς. το κινέζικο σύστημα δηλαδή είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στο IFRS και εμείς τους θεωρούμε πραγματικά μέλη της οικογένειας και άλλωστε συμμετέχουν και σημαντικά στον προπολογισμό μα Είναι πολύ πιο εμπλεκόμενοι οι Κινέζοι ε, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς. Τώρα για τα, ψηφι... για τα ε, ψηφιακά νομίσματα, οικονομικά νομίσματα. Όπως ίσως γνωρίζετε, για να αναπτυχθεί ένα πρότυπο χρειάζεται περίπου 5 χρόνια. Και θεωρώ ότι μέχρι ότου τελειώσουμε την προσπάθεια αυτή, ίσως να έχουν εξαφανιστεί τελείω τα εικονικά νομίσματα. Και φαίνεται αυτή να είναι εξέλιξη για την ώρα. Εξάλλου, βάζοντας, δημιουργώντας ένα πρότυπο, στην ουσία νομιμοποιείται την αγορά. Ενώ η αγορά των οικονομικών νομισμάτων έχει πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Δεν είναι καθόλου σωστά. Και γι' αυτό διστάζουμε. Τέλος, αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε είναι να μας δώσει η Interpretation Committee κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα εικονικά νομίσματα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Δίνουμε μια γενική κατεύθυνση. Τώρα δεν είμαι βέβαιος αν κατάλαβα απολύτως την ε, μεσαία σας ερώτηση για top line και bottom line, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Εμείς φτιάχνουμε τώρα ένα πρότυπο για income statement, για ε, δηλώσεις εισοδήματος δηλαδή που είναι πολύ πιο λεπτομερές ώστε να αντιμετωπίσουμε κενά τα οποία υπάρχουν από ανταχού του κόσμου. Ε, ε, αυτό νομίζω ότι μπορεί να είναι η απάντηση στην ερώτησή αλλά ίσω και να μην, την εννοεί, να μην την κατανόησα σωστά. Τώρα, ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Κύριε Ουρτασούν, όχι. Δεν βλέπω μέλη άλλων πολιτικών ομάδων. Αν δεν έχετε ερωτήσεις στο σύστημα Catch νομίζω τότε ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτηση με τους δύο προσκεκλημένους μας, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερως για, για την ε, πολύ ζωντανή ανταλλαγή απόψεων που μου φάνηκε και πολύ χρήσιμη. Όπως είπα, θα συνεχίσουμε. Είμαι άλλωστε βέβαιος ότι η Νομισματική Επιτροπή, όσοι εξημών θα παραμείνουμε εδώ, Ασφαλώς θα συνεχίσουμε τον διάλογο μαζί σας και όπως είδαμε σήμερα υπάρχουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα τα οποία θα χρειαστεί να συζητήσουμε Η συζήτηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη διότι υπάρχουν και κάποιες διαφορές, για παράδειγμα για την αναχώρα ε, υποβολή εκθέσεων. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συνεργασία σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Dear colleagues. Ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Dear colleagues, may I ask you to take seat. Σας παρακαλώ να καθίσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και όσοι παρακαλώ, όσοι επιθυμούν να συνομιλήσουν, ας περάσουν έξω. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Και αρχίζουμε με την λίστα ακροάσεων. Πρώτος δε, πρώτη μάλλον, είναι η δημόσια ακρόαση με τον προτινόμενο υποψήφιο για την θέση πλήρους μέλους του Single Resolution Board. Έχω τον κύριο Λαβιόλα δίπλα μου. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Λαβιόλα, ως γνωρίζετε, εξετάζουμε στην ακρόαση αυτή τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πλήρωση κενών θέσεων στον ενίο μηχανισμό εξηγιάνσεων, διότι παρατήθηκε ο κύριος Γκράντε. Εύχομαι το καλό ορίσατε στον κύριο Λαβιόλα που είναι ο υποψήφιος που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, τα μέλη της ε, Ομάδα ε, που ασχολούνται με, τις, ε, με τα τραπεζικά κτλ. Συναντήθηκαν ήδη με τον κύριο Λαβιόλα στι 15 Ιανουαρίου, όταν προτάθηκε η υποψηφιότητα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται τώρα για τη δεύτερη φάση με δημόσια ακρόαση, που παίζει σημαντικό ρόλο για τα μέλη του ERSB και για τη λογοδοσία των μελών, για τις αποφάσεις τους σχετικά με την έγκριση ή μη του υποψηφίου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Σε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε λάβει νομίζω και αντίγραφα του βιογραφικού του κ. Λαβιόλα, στον οποίο θα δώσω αμέσως τον λόγο για να προβεί σε μια εισαγωγική τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ στην ακρόαση αυτή για να οριστώ ως μέλος του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης. Θέλω να σας αναφέρω την εμπειρία μου στη δουλειά μου και να σας πω γιατί είμαι υποψήφιος και τι θα προσφέρω στο Συμβούλιο αυτό. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 ήμουνα στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουλέψω εκεί και συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις, στα διάφορα στάδια και γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα τραπεζικά και με τα χρηματοπιστωτικά. Πριν έρθω στις Βρυξέλλες, όλη μου τη ζωή ασχολήθηκα λίγο πολύ με θέματα εξυγίανσης και εποπτείας τραπεζών. Ήμουνα μέλος συμμέτοχος διεθνών εποπτικών ομάδων μέχρι το 2012 από το 2001. Μετά από έξι χρόνια διαπραγματεύσεων τεχνικών και πολιτικών στο Συμβούλιο, ευχαρίστως θα προσφέρω τη δικιά μου συνεισφορά στην διαχείριση. Η δημιουργία ενό πλησίου εξυγίανση τραπεζών στην Ευρώπη είναι κάτι πολύ σύνθετο και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε, το 2000, ε, ξεκίνησε από το τίποτα, είναι πολύ σημαντικό το τι έχει πετύχει μέχρι τώρα. Βέβαια πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο. Για παράδειγμα, το έργο συνεχίζεται για εξυγένση όλων των τραπεζών στα πλαίσια του Ενίου Συμβουλίου Θέλουμε να βασιστούμε στη δουλειά που έχει ήδη γίνει, αλλά βέβαια πρέπει και να αξιολογήσουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Οι εξελίξεις MRL και οι στόχοι που παγιώνονται σε κάθε επίπεδο μας οδηγούν σε μια νέα νομοθεσία για το MRL και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα επιπλέον στόχος θα είναι αναλυτικό και πολιτικό έργο για να μην υπάρχουν πια προβλήματα. Θα δουλέψουμε και θα συνεργαστούμε περισσότερο με τις αρχές, τις νομισματικές και τις οικονομικές, όχι μόνο στις χώρες Ευρωζώνης, αλλά και εκτός αυτής. Και βέβαια το τι θα γίνει μετά το Brexit παίζει εδώ κάποιο ρόλο. Τέλος, η εμπειρία που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας οδηγεί να προβληματιστούμε για βελτίωση του πλαισίου. Η διάθεση ρευστότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο μηχανισμού αρκετά ευέλικτου και με το κατάλληλο μέγεθο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μα για την εξυγίανση των τραπεζών. Που σημαίνει ότι έτσι θα μπούμε ε, στο ίδιο επίπεδο με τι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της διάσκεψης του καλοκαιριού μας πέρασε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κληθεί να στηρίξει την Επιτροπή και τις χώρες μέλη για να ε, προλάβουμε τις επιπτώσεις από ένα backstop και θα δημιουργήσουμε και το σχέδιο για τις εγγύσεις καταθέσεων. Δεδομένου βέβαια ότι η εξυγίανση θα εφαρμοστεί μόνο σε ένα μέρος των τραπεζών, ε, το καθεστώς έλλειψης ρευστότητας για τις τράπεζες αποτελεί ένα πρόβλημα. Υπάρχουν διαφορές στις χώρες της Ευρωζώνης, διαφορετικά καθεστώτα, που σημαίνει ότι η αξιολόγηση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και δεν μπορεί να διευκολυνθεί το έργο. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε στην Ευρώπη να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό καθεστώ για μικρού μεγέθου και μεσαίου μεγέθου τράπεζε που δεν υποβάλλονται στο σχέδιο εξυγίανση. Να δημιουργηθεί ένα διοικητικό μέσο, για παράδειγμα, όπω προτείνει και το Δουνουτού. Τώρα θα αποτελέσει ένα παράθυρο ευκαιρία πολύ πιθανόν γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να βοηθήσει με συμβουλέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πού πρέπει να υπάρχει η εναρμόνιση και με ποιο τρόπο. Οπότε αυτό θα είναι υποφελέ δηλαδή. Η ανάπτυξη πολιτικής και συντονισμού επίσης θα συμμετέχει για το έργο αυτό όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και ανάληψη ευθύνων στο Συμβούλιο για την δημιουργία σχεδίων εξυγίνησης μέσα σε το πολιετές προγραμματισμό, στο συντονισμό επίσης εκθέσεων αξιολόγησης, όπως επίσης και υπέρ της συνεργασίας με εθνικές αρχές. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα με τις αρχές ακόμα και σε τρίτες χώρες. Επ' αυτού λοιπόν πιστεύω ότι διαχειριστικές ικανότητες είναι κάτι πολύ σημαντικό και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις εμπειρίες που έχω συλλέξει κατά το παρελθόν. Όσον αφορά την πολιτική κρίση, επίσης η συνεργασία ε, σε περίπτωση κρίσεων, ηγεσία κτλ. βοηθάει. Τα έχω κάνει κατά τη σταδιοδρομία μου. Έχω συλλέξει ε, τεχνική γνώση που επίσης θα μπορέσει να χρησιμεύσει πολύ. Συχνά ήμουν πρόεδρος σε διάφορες επιτροπές και άρα έχω τα προσόντα για να αντιμετωπίζω ευαίσθητα ζητήματα που δημιουργούν κρίσεις και διαμάχες με εθνικές αρχές. Στο ιδιωτικό τομέα τώρα είχα ε, επίση αρμοδιότητες. Η διαφάνεια για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα κατακλείδι. Έχοντας διαπραγματευτεί ε, το σχέδιο για την Κεφαλιακή Ένωση, εφόσον ε, εγκριθώ στον ορισμό μου, θα μπορέσω να βοηθήσω την υλοποίησή του και θα συνεισφάλω στην οτροπία την ευρωπαϊκή για αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι μια τραπεζική ένωση καλά οργανωμένη και που λειτουργεί με διαφάνεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όσο σημαντικό ήταν και το νέο νόμισμα. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαβιόλα. Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις των μελών. Πρώτος ο κύριος Φέρμπερ. Θα σας τα πω στα γερμανικά φορές τα ακουστικά σας, σας παρακαλώ κύριε Βιόλα, διότι έχουμε και την ε, διερμηνία όσο αντιλαμβάνεστε. Αυτή είναι η διαφορά άλλωστε σε σχέση με τις άτυπες συναντήσεις. Μιλώ γερμανικά. Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε τι σας λέω μέσω της διερμηνίας. Ακούω τώρα. Ένα, δύο, τρία. Περιμένω να μου απαντήσετε αν ακούτε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 Ça Μπορώ να μιλήσω γερμανικά τώρα, ρωτάω και ο Φέρμπερ. Θαυμάσια. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαβιόλα. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει μαζί σα σήμερα. Πολύ συγκεκριμένα, του τελευταίου μήνε υπήρξαν περιπτώσει όπου αναγκάστηκαν να διασωθούν τράπεζε με χρήματα φορολογουμένων. Όπω η Banca Popolare di Vicenza, η Banca Carice και άλλε Ιταλικέ τράπεζε, δηλαδή. Η υπόσχεση τη τραπεζική Ένωση, ωστόσο ήταν ότι ο φορολογούμενος δεν θα κληθεί πλέον να διασώσει τράπεζε. Ωστόσο τώρα δημιουργείται η εντύπωση ότι σε ορισμένε περιπτώσει καταστρατηγείται τουλάχιστον το πνεύμα του καθεστώτος αυτού. Πώ αξιολογείται τι περιπτώσει αυτέ, Υπάρχουν ασυνέπειε σε ό,τι ε, αφορά την ε, τήρηση των προβλέψεων του καθεστώτος εξηγιάνσεως ή πού εντοπίζονται τα προβλήματα. Δεύτερη ερώτηση. Πού βλέπετε να εντοπίζονται τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την σταθερότητα του τραπεζικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις και πώς πρέπει να γίνουν αυτές. Αυτά πολύ σύντομα είναι οι δύο ερωτήσεις αυτές μάλλον που εντοπιζονται τα προβληματα δευτερη ερωτηση που βλεπετε να εντοπιζονται τωρα τα μεγαλυτερα προβληματα σε οτι αφορα την σταθεροτητα του τραπεζικου τομεα στην ευρωπαικη ενωση που πρεπει να επελθουν βελτιωσει και πως πρεπει να γινουν αυτες αυτα πολυ συντομα ειναι οι δυο ερωτησει αυτε μαλλον που ειχα προ εσά. So, let me recap the questions if I understood correctly. Ανακεφαλαιώσω ε, για να δω αν κατάλαβα καλά. Ε, νομίζω ζητήσατε στην αρχή να καταλάβετε εάν στις περιπτώσεις διάσωσης ή τέλος πάντων στις κρίσεις υπήρχε παραβίαση ή κάποια, κάποιος κλειδονισμός στο πλαίσιο διάσωσης για την Τραπεζική Ένωση όπως προβλέπετε. Ε, Είχαμε αρκετές εμπειρίες περιπτώσεων κρίσης, τριγμών Ευρώπη, στην Ευρώπη που απέτησαν διάσωση. Δηλαδή τη δική μας την ε, παρέμβαση του SRB, ε, ε, του Banco Popular, και κάποιες φορές ανακεφαλαιοποίηση ή ρευστοποίηση. Όπω στην περίπτωση τη Τράπεζα Βένετο, του Βένετο. Ε, σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, οι κανονισμοί και οι κανόνε έγιναν πλήρω σεβαστοί. Δεν υπάρχει θέμα οποιασδήποτε παραβίαση, παράβαση και ούτω καθεξής. Αυτό που υπενήσαστε εσεί είναι ότι το πνεύμα ίσως ήταν ε, διαφορετικό σε σχέση με αυτό που προβλέπετε από τους κανόνες. Καταρχάς υπήρχαν θέματα αγορά. που ε, όπως η νομοθεσία είναι πολύ φρέσκια, ήταν ε, σαν δοκιμές αυτές οι περιπτώσεις οι πρώτες. Να θα δώσω ένα παράδειγμα, στην περίπτωση του Banco, του Banco Veneto. Ε, υπήρχε διαφορά μεταξύ της αξιολόγησης του SRB και των διεθνών και ευρωπαϊκών χρηματαγορών για το πώς πήγαινε η τράπεζα, καθώς και την αποτίμηση της εθνικής των εθνικών αρχών για την οικονομική σταθερότητα και την ε, δυνατότητα αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τι τοπικέ αρχέ. Είναι σίγουρα αυτό απολύτω συμβατό με την νομοθεσία, την νομοθεσία που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα το αν μπορούσαμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά ή αν μπορούσαμε να, επανεξ, να επαναξιολογήσουμε τις διαφορές αυτές στην ε, αποτίμηση του δημόσιου συμφέροντος στην ε, περίπτωση αυτή. Εδώ υπάρχει δυνατότητα να το σκεφτούμε. Κάτι άλλο που ε, αναφέρθηκε σε αυτή την περίπτωση είναι η διαφορά μεταξύ της ιεράρχησης των ε, πιστωτών, ποιος πληρώνει το λογαριασμό στην περίπτωση της διάσωσης και ποιος στην περίπτωση της ρευτοποίησης, της πώλησης δηλαδή. Ε, θα μπορούσαν οι πιστωτέ που είναι senior, τέλο πάντων αυτοί που έχουν τι περισσότερε δυνατότητε να έχουν προσελκυστεί, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε για άλλου λόγου. Πρέπει να το σκεφτούμε, διότι σίγουρα οι δύο τομείς θα μπορούσαν να συνδυαστούν, αλλά ο πρόεδρος του SRB και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουν στηρίξει αυτή τη γραμμή. Πρέπει να παραδεχτώ ότι κι άλλα έχουν φανεί από την πρόσφατη κρίση. Στον Banco Popular, ας πούμε, διαπιστώσαμε ότι αυτό που μας λείπει είναι ένα πλαίσιο χρηματοδότησης σε περίπτωση διάσωσης. Κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό, ακόμη και αν μια διάσωση αγορά, αγορά γίνει σωστά. Η τράπεζα θέλει χρόνο για να ανακτήσει τη φήμη της στην αγορά και την εμπιστοσύνη των πελατών. Υπάρχουν παράπλευρες απώλειες το backstop και οι πόροι μας για τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες δεν είναι ακόμα αρκετά. Θα χρειαστεί και κάποιος άλλος ε, φορέας να πάρει μέρος, ίσως μια κεντρική τράπεζα. Ούτε αυτό όμως είναι εγγύηση και τώρα το ερώτημα είναι ποιος θα προσφέρει τις εγγύησεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα. Νομίζω οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν κάνει πολλά για την κρίση ως προς την αύξηση του κεφαλαίου και των επιπέδων ρευστότητας. Σίγουρα είναι πιο ανθεκτικές και πιο σταθερές σε σχέση με την αρχή της κρίσης. Αυτό που εγώ βλέπω ως πρόβλημα είναι να συνεχιστεί η δουλειά στα MPL. Ε, που έχει ξεκινήσει από την αρχή της κρίσης να μελετάτε, όπως στην Ιταλία το 2015, αλλά έχουν προκύψει και άλλα θέματα. Φταίει και η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο εμπορικός προστατευτισμό που έχει αναδυθεί. Έχουμε λοιπόν δυσκολίες στην αγορά. Χρηματοδότησης κυρίως. Σίγουρα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις, ιδίως για την κερδοφορία των τραπεζών και την αξιολόγηση των τραπεζών, ιδίω την υπερβολική δυνατότητα που έχουν κάποιε φορέ. Πιστεύω άρα ότι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των τραπεζικών μοντέλων και των επιχειρηματικών μοντέλων είναι προαπαιτούμενο ώστε να είναι οι τράπεζε βιώσιμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε, Περβάνη Μπερέ. Όχι, όχι. Ε, κυρία Βίντερ. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, ναι. Και εγώ θέλω να μιλήσω γερμανικά, αν δεν έχετε αντίρρηση, αν παρακολουθεί τη διερμηνία, κύριε Λαβιόλα. Ευχαριστώ, κύριε Λαβιόλα, λοιπόν, για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σας σχετικά με τα όσα ήδη έχουν επιτευχθεί για την διασφάλιση των τραπεζών, διότι αν εξετάσει κανείς τα τελευταία χρόνια, προ πέντε ετών αντιμετωπίζαμε πάλι ευρωεκλογές και τα συζητούσαμε τέτοια πράγματα τότε όπως και τώρα. Ωστόσο έχω κάποιες ερωτήσεις. Αφενός μια γενική ερώτηση, αν δείτε την ασφάλεια της Ευρωζώνης, με, μπορείτε να με παρακολουθήσετε, έχετε τη μετάφραση. Από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν αρχίσει και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ποιες έχουν προτεραιότητα κατά τη γνώμη σας Δεύτερο, κάπως πιο εξειδικευμένο ερώτημα. Μιλήσατε για μηχανισμούς αφαιρεγγιότητας. Εγώ ε, έχω διαδεχθεί τον κύριο Βάιτζέκερ και έχω αναλάβει και μια εισήγησή του για Case Winburn σχετικά με νομοθέτημα του Κοινοβουλίου και, των, ε, και του Συμβουλίου για ε, εξυγιάνσεις κεντρικών μερών. Το ερώτημά μου προς εσάς είναι, διότι ε, μιλήσατε κι εσείς για τον μηχανισμό αφαιρεγγιοτήτων, αν μπορεί και πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός αντισυμβαλωμένων για την εξυγίανση αντισυμβαλωμένων των τραπεζών, ώστε να αποφευθεί ένα ενδεχόμενο, μια ενδεχόμενη ε, άτακτη κατάρρευση τραπεζών. Ξέρω ότι ε, μάλλον έχω ε, την κυρία Σουίνμπερν με την οποία συνεργάζομαι και θέλουμε να φέρουμε την έκθεση στην Ολομέλεια. Η έκθεση αυτή έχει συζητηθεί ήδη εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών. Ήθελα να ακούσω την απάντησή σας γιατί μιλήσατε ήδη για τους μηχανισμούς αντιμετώπισης αφαιρεγγιωτήτων. Ε, ευχαριστώ πιο επίγουσες μεταρρυθμίσεις της Ευρωζώνης. Βεβαίως μιλώ μόνο για τα νομισματικά, διότι εκεί ασχολούμαι. Βεβαίως η Τραπεζική Ένωση ξεκίνησε μισό επιτεύχθηκε αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Αυτό που χρειαζόμαστε και νομίζω τα γνωρίζουν όλοι αυτά, Single Resolution Fund, ενίο ταμείο εξηγιάνσεων, μηχανισμός ε, κοινής διαχειρίσεως και σύστημα εξασφάλισης των αποταμιέσεων. Αυτό των καταθέσεων δηλαδή. Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως χώρας από την οποία προέρχονται. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια που δεν έχουν επιτευχθεί εμποδίζουν διότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος ανάμεσα στους δύο παράγοντες που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και στην συμπεριφορά ring fencing δηλαδή διασφάλισης των ε, κεντρικών ε, αρχών. για την διαχείριση ταμείων για τις διαμεθοριακές επιχειρήσεις και παρεμποδίζει αυτή η υπόθεση και τις διαμεθοριακές συγχωνεύσεις που θα ήταν σημαντικές για να μειωθεί το υπερβάλλον δυναμικό που ε, έχουν ορισμένε τράπεζε σήμερα στην Ευρώπη. Άρα χρειαζόμαστε ενίο μηχανισμό εξηγιάνσεων το και αυτό που είπα η χρηματοδότηση των εξηγιάνσεων. Γιατί οι εξηγιάνσεις πρέπει να είναι βέβαια αξιόπιστες. Μίλησα για τον μηχανισμό αφαιρεγγιοτήτων. Τράπεζες που δεν πηγαίνουν στην εξηγένση αυτές αφορούνται εδώ. Είναι σημαντικό και έχει τονιστεί και φάνηκε καθαρά και στην κρίση της EBLV, της, Λατινική, της ε, Η, υπήρχε η Τράπεζα Χαρτοφυλακίου και η θηγατρική της στο Λουξεμβούργο. Έγινε αφενός αυτοεξυγένση από το Συμβούλιο της Τράπεζας και από την άλλη μεριά όμως για την άλλη για τη θεατρική υπήρξε μονάχα πάψη πληρωμών, διότι η κρίση τους ήταν διαφορετική από αυτή που θα είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και εμεί ω ESRB. Αυτά όμως ήταν και αναμενόμενα, αναμενόμενα θέματα ε, Αυτά υπονομεύουν την ε, εφαρμογή των αρχών για διαμεθοριακού ομίλου. Δηλαδή τελικώ υπάρχει διαφορετική μεταχείριση που επιφυλάσσεται για δύο τράπεζε του ίδιου ομίλου. Πρέπει ε, να εξεταστεί το δημόσιο συμφέρον, διότι εάν δεν πρόκειται για εξυγίανση, τότε σημαίνει αφαιρεγγιότητα. Μπορεί όμως εκεί η απόφαση τελικώ να έχει διαφορετικά αποτελέσματα στι δύο χώρε που αφορούνται τώρα για την έκθεση για την ολοκλήρωση των CCP και την έκθεση κυρία Σουίνμπερν. Οφείλω να πω ότι στο ESRB, στο Συμβούλιο δηλαδή, δεν έχει συζητηθεί το θέμα αυτό εξ όσων γνωρίζω. Είναι αληθές επίσης, υπάρχει μια τάση μεταξύ των, και μάλλον μια ένταση μεταξύ των κεντρικών αρχών που θεωρούν ότι η διαχείριση CCP των πτωχεύσεων μπορεί να κέντρο, να γίνει κεντρικά. Όσο δηλαδή η δημοσιονομική ευθύνη παραμένει εθνική, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο στην πορεία αυτή, θα πρέπει να βρούμε μια εφαρμόσιμη λύση για το πρόβλημα αυτό. Διότι στην περίπτωση του Συμβουλίου έχουμε συγκεντρώσει τις αποφάσεις, αλλά τις έχουμε συγκεντρώσει και τα κονδύλια. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Τρεμόζα. Πρώτα εσεί όχι. Με ποιο Τρεμόζα. Hello, ok. okay. Grazie Presidente. Buongiorno, benvenuto signore Laviola. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Λαβιόλα και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρεις ερωτήσεις έχω σύντομα. Πρώτον, το πολύ μεγάλη για να κλείσει μια τράπεζα. Κατά τη γνώμη σας τι θα πει πολύ μεγάλη, πόσο. Ξέρετε στην Αμερική 70 τράπεζες ε, αναγκάστηκαν να κλείσουν με την κρίση και τα χρήματα πήγανε για τις τράπεζες που θα μπορούσαν να αγοραστούν. Ποια είναι η γνώμη σας. Δεύτερον, ποια είναι η γνώμη σας για τη συγκέντρωση των τραπεζών. Στην Ευρώπη υπάρχουν δύο τάσεις. Στην Νότια Ευρώπη ε, η προτίμηση είναι να υπάρχουν τρεις, τέσσερις, πέντε ε, μεγάλες εθνικές. Δεν υπάρχει πολύ περιθώριο για αποταμιευτικές τράπεζες, ενώ αλλού συνδυάζονται και υπάρχουν πάρα πολλέ μικρές περιφερειακές τράπεζες. Ποια είναι η γνώμη σα. Και τρίτον, το ελεγκτικό συνέδριο, το ευρωπαϊκό, έκανε μία ανακοίνωση για τις ε, αποκαλύψεις για τον ECA. Εσείς πώς βλέπετε τις βελτιώσεις όσον αφορά τη λογοδοσία του ε, συμβουλίου του δικού σας. Ευχαριστώ. Όταν μια τράπεζα είναι πολύ μεγάλη για να κλείσει, πότε. Ναι, πολύ δύσκολη η ερώτησή σας αυτή και δεν νομίζω ότι έχει κανείς μια ακριβή και σωστή απάντηση. Εξαρτάται. Αυτό όμω που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτά που γίνανε στην ε, χρηματοπιστωτική κρίση όπου κλήθηκαν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν το λογαριασμό, δεν θα έπρεπε να επανεληφθεί. Οπότε το πλαίσιο της εξυγένσης άλλαξε. Πρώτα απ' όλα υπήρξε το Διεθνές ε, Συμβούλιο Σταθερότητας και μετά με όλες τις ιδιαιτερότητες έγινε κάτι και στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ποτέ πια μια τράπεζα που να είναι πολύ μεγάλη και άρα να πρέπει να διασωθεί και να μην κλείσει. Ε, δεν ξέρω τι να σας πω. Σίγουρα έχουμε πολλές ρήτρε ασφάλειας τώρα. Έχουμε τον Μπέιλιν, έχουμε τα επίπεδα των ελάχιστων απαιτήσεων ε, ιδίων πόρων για τις τράπεζες, το ΜΡΕΛ. Πάντως, όταν ε, ε, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το Συμβούλιο Εξυγένσης, είναι ακριβώς για να αντιμετωπίζονται τα πολλαπλά σοκ και να μην υπάρχει το πρόβλημα που είχαμε με την κρίση, κυρίως για τις μικρές, τις μεσαίες Γι' αυτό όμως ακριβώς και η παρέμβαση των δημοσίων αρχών είναι κάτι καθοριστικό στα πλαίσια της οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών. Τώρα υπάρχει το μοντέλο, είπατε, που ανθίζει στο νότο για τις τράπεζες. Και ρωτάτε τη γνώμη μου. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι οι ρυθμιστικές αρχές, οι δημόσιες αρχές μιας χώρας που αποφασίζει ποιο μοντέλο θα αναπτυχθεί. Οι τράπεζες είναι επιχειρηματίες. Πρέπει ο ιδιοκτήτης τους να αποφασίσει πρώτα απ' όλα. Και μετά βέβαια ανάλογα με το τι γίνεται με τις δυνάμεις της αγοράς, τι γίνεται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ανάλογα κυρίως στην Νότια Ευρώπη που χτυπήθηκε πάρα πολύ από τη χρηματοπιστωτική κρίση, αργότερα αλλά πάρα πολύ, εκεί υπάρχει τάση συγκέντρωσης. Αναδύθηκε αυτή η τάση. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση των αποταμιεύσεων και να περιοριστεί σε μερικές περιπτώσεις η υπερβολική ικανότητα. Τώρα να συνεχίσουμε να έχουμε ένα πλήρες ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου να υπάρχει κεφαλαϊκή ρευστοποίηση κτλ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο τις ε, διαφορές ανάμεσα στο τραπεζικό μοντέλο της μίας ή της άλλης χώρας. Οι τράπεζες θα είναι ευρωπαϊκές, τελείωσε. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είναι χρήσιμες οι μικρές τράπεζες, κάθε άλλο. Οι μικρές τράπεζες μπορούν να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν τους πιο μικρούς πελάτες τους. τα συμφέροντα και αυτών που μπορεί να είναι λίγα, όχι τόσο σημαντικά, πρέπει να εξυπηρετούνται. Οπότε όταν συζητάμε το μέγεθος και το είδος προσφοράς, όλα είναι αναγκαία στην πραγματική οικονομία παντού στην Ευρώπη. Τώρα για το ελεγκτικό συνέδριο και την έκθεσή του για το RSB. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστηματικού Κινδύνου. Διάβασα και εγώ την έκθεση, αλλά από κάτι καταλαβαίνω εγώ, Ευρω... είπε ότι υπάρχουν πληροφορίες για τις οποίες χρειάζεται άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν ε, αποκαλυφθούν, πριν κυκλοφορήσουν. Οπότε από αυτού δεν μπορώ να πω περισσότερα από αυτά που διάβασα κι εγώ στην έκθεση και από την απάντηση του ESRB. Όσον αφορά τώρα την βελτίωση ε, της ε, ενημέρωσης, πάλι κοιτώντα απ' έξω και με κάθε σεβασμό για τα όσα έχουν ήδη γίνει και βελτιωθεί όλα αυτά τα χρόνια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ξεκινώντας από την ιστοσελίδα και ίσως βέβαια από κάποια καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ουρτασούν τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Λαβιόλα. Έχω μερικές ερωτήσεις, επιτρέψτε μου. Πρώτα απ' όλα, και εσείς στην αρχή αναφερθήκατε στο πρόβλημα της προετοιμασίας του σχεδίου εξυγένσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε αργήσει. Όμως θα ήθελα να ξέρω τώρα ποια είναι η δικιά σας ιδέα, πώς μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία και πώς πιστεύετε ότι πρέπει να δουλέψει το ESRB προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στη διαδικασία. Δεύτερον, για την προστασία των καταναλωτών και για την πώληση μετοχών MRL. Εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορούν να προστατευτούν οι μικροί αποταμιευτές. Ήδη έχουμε εισαγάγει κάποια νέα μέτρα. Ζητούμε για παράδειγμα δοκιμές καταλληλότητας ή βάζουμε κάποιο όριο, κάποια οροφή. Αλλά κάτι το οποίο παραμένει ανοιχτό είναι τι γίνεται αν ένα προϊόν είναι μεν επιλεκτικό, για το MRL, αλλά τελικά δεν πουληθεί. Θα ήθελα να ξέρω να μου πείτε εσείς πώς μπορούν να προστατευτούν οι άνθρωποι από τέτοιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Τώρα, πώς να επιταχύνουμε, λέτε, την διαδικασία όσον αφορά τα σχέδια εξηγένσης. Από ό,τι και πάλι έχω διαβάσει και κρίνοντας απ' έξω τα πράγματα, για φέτος και το πολιτές πρόγραμμα, θα ολοκληρωθεί το 2020. Στο τέλος δηλαδή ε, της, του 20 ε, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για το ενίο Συμβούλιο Εξυγένσης. Μέχρι τώρα έκανα άλλη δουλειά, οπότε δεν ε, μπορώ να σας τα πω από μέσα. Είναι σημαντικό πάντως η δουλειά να γίνει τώρα και πλησιάζουμε στο τέλος για τα λιγότερο σημαντικά όργανα, μία τράπεζες κτλ. Έχουν ολοκληρωθεί κάποια σχέδια, κάποια παραμένουν. Πρέπει να γίνει όμως για όλες τις τράπεζες, αυτό είναι αλήθεια. Για τις άλλες τράπεζες Τώρα που έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα, νομίζω ότι το σχέδιο εξηγένση είναι ζωντανό οργανισμό. Έτσι, δεν είναι ότι τον αφήνει στην πάντα. Πρέπει να συνεχίσει η ενημέρωσή του, γιατί προκύπτουν νέα προβλήματα, νέοι κίνδυνοι, νέα business models. Οπότε εδώ πιστεύω ότι αυτό στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί το Συμβούλιο εξηγένση είναι να προβάλλει το έργο του, κάτι το οποίο δεν γίνεται πάντα συστηματικά, να γίνει παρετέρω αξιολόγηση, κάποια έχει ήδη γίνει, αλλά να δούμε και την καταλληλότητα της λειτουργίας ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξηγένσης και τις εθνικές αντίστοιχες αρχές και αυτό να γίνει και με τις αρχές εκτός Κεφαλιακής Ένωσης και μετά να καταλήξουμε σε μια ασφαλή πολιτική MRL, ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, και η νομοθεσία να βοηθήσει ώστε να υπάρξει κατάλληλη προστασία, χωρίς όμως η υπερβολική παρέμβαση στην αγορά. Γιατί αυτό θα ήταν δύσκολο. Στην περίπτωση του mis-selling, έχετε κι εσείς αναφέρει συγκεκριμένα περιπτώσεις, είναι σαφείς οι κανόνες που ισχύουν. ο μικρός ε, επενδυτής πρέπει να περάσει το πρώτο τεστ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι με την πρώτη προσπάθεια δεν ήταν αρκετά σαφή τα πράγματα. Οι επόπτες ε, στη συνέχεια ήταν σαφέστεροι και στη χώρα μου για το τι πρέπει να κάνει η τράπεζα, τι πρέπει να προσέξει, αλλά τι πρέπει να προσέξει και ο επενδυτής τα ξέρει πλέον σήμερα. Ε, το τεστ καταλληλότητας είναι ζωτική σημασίας. Έχουμε πει ότι δεν μπορεί ένας μικρός χρήστης να απαγορευτεί να γραφτεί σε ένα πρόγραμμα τέτοιο. Αλλά θα έπρεπε οι αρχές να βοηθούν. Τώρα αν γίνει αυτό που περιγράψατε κι εσείς, πρέπει να εκτιμάται κατά περίπτωση. Το μη selling δεν είναι ότι κάποιος πρέπει να αποφεύγει στη συνέχεια το αίτημα για bail Σίγουρα όμως πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση και να υπάρχει μια διέξοδο, αν αποδειχθεί ότι όντως έχει γίνει μη selling. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να είναι κανείς εδώ από την ΚΟΕ, ούτε για τις άλλες ομάδες. Οπότε, εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, κάτι να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Α, Περβάνης, έχετε το λόγο. Με συγχωρείτε, αλλά ξεχάστηκα. Εάν κοιτάξει κανείς τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, μπορεί να σκεφτεί ότι το backstop του Ταμείου Διάσωσης θα ενταχθεί στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Σταθερότητας. Αυτό όμως με οδηγεί να σας θέσω ένα ευρύτερο ερώτημα για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ένα εργαλείο διακυβερνητικό προς στιγμή. Το Ταμείο Διάσωσης που είναι κοινοτικό κάπως θα ε, για να το πω έτσι, από την ένταξη ενός διακυβερνητικού μηχανισμού. Πιστεύετε ότι μακροπρόθεσμα θα πρέπει να φύγουμε από τη λογική των ε, διακυβερνητικών μηχανισμών ώστε να είναι κοινοτικά όλα αυτά όπως έχει ζητήσει από την αρχική επιμένει να ζητά το Κοινοβούλιο Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Παρόλο που σας κατάλαβα. Ναι, δεν χρειάζομαι τα ακουστικά, μπερδεύτηκα. Θα απαντήσω αγγλικά. Ναι, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα είναι διακυβερνητικό. Ξέρουμε γιατί δημιουργήθηκε και το Ταμείο είναι ευρωπαϊκό λέτε ότι εάν ο μηχανισμός τελικά διαχειρίζεται το backstop θα υπάρχει κάποιο είδους ε, επιμόλυνση γιατί ο κανόνας είναι η ομοφωνία στη μία περίπτωση, ενώ σε περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης και το καθεξής θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις διακυβέρνησης που ακόμα δεν έχουν οριστεί. Αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συνταγματικές απαιτήσει και το καθεξής. και επίσης να ε, γίνεται σεβαστή και το επίγον της απόφασης. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ε, συνολική της μεταρρύθμιση για την Ευρωζώνη, υπήρχε η πρόθεση σιγά σιγά ο μηχανισμός σταθερότητας να μετατραπεί σε ευρωπαϊκό από διακυβερνητικό. Άρα εδώ το θέμα, μακροπρόθεσμα, μπορεί να είναι ε, έτσι ως τελική λύση. Διότι αν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί είναι μετελείς και αν μια μέρα το ε, είναι ένα σύνολο εθνικών αποφάσεων, δεν καταφέρνουμε τίποτα πρέπει να έρθουν σε κεντρικό επίπεδο οι ευθύνε και τα ταμεία. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει ε, συμβατότητα μεταξύ του τι συμβαίνει αν μια τράπεζα πτωχεύσει και ε, πρέπει να απολυθεί, οπότε τη λυπητέρη την πληρώνει ένα κάποιο και τι γίνεται με το αν υπάρχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Αν δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ε, λόγω του μεγέθου των ποσών και του ευρωπαϊκού μηχανισμού, εάν όλα ήταν σε κεντρικό επίπεδο. Θα ήταν πιο εύκολο για κυβέρνηση, πιστεύω εγώ. Ε, αυτή είναι η δική μου απάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα όχι βραχυπρόθεσμα, ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα όμως. Σίγουρα θα το επιθυμούσε το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψεις όμω ίσω στο Eurogroup. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συναλλαγή, για την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε που είχαμε. Dear colleagues. και αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε στο υπαριθμό 10 της ημερησία διατάξεως μας περί διορισμού μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και απευθύνω το καλώ ορίσατε στον ε, Ιρλανδό Κεντρικό Τραπεζίτη κύριο Λέιν. Καλώς ήρθατε, με χαρά μας σας ε, βλέπουμε εδώ και ω γνωρίζετε το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ αποφάσισε στις 12 Φεβρουαρίου να προτείνει την υποψηφιότητα του κυρίου Λέιν ως Chief Economist για το Συμβούλιο της, Κεντρικής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα αντικαταστήσει τον κύριο Πάτ από την 1η Ιουνίου 2019 για 8 χρόνια. Γνωρίζετε και δεν είναι άλλωστε και κανένα μυστικό ότι είχαμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε άτυπη ανταλλαγή απόψεων σε προηγούμενη ευκαιρία με τον κύριο Λέιν και, και το Κοινοβούλιο απεκόμισε εξαιρετική εντύπωση σχετικά με τα προσόντα του κύριου Λέιν. Είναι λοιπόν μεγάλη ευχαρίστηση για μένα και για όλους μας που έχει προταθεί η υποψηφιότητά σας από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Και Ε, Ευχαριστώ. Διεξάγουμε και την επίσημη πλέον άκουραση μαζί σας. Πρόκειται για διαδικασία διαβουλεύσεως και θα προχωρήσουμε με μια πρώτη τοποθέτηση δική σας και μετά με ε, ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, χαίρομαι πολύ που έχω τη δυνατότητα να εμφανιστώ σήμερα μπροστά και ιδίως σε ό,τι αφορά το, τον ρόλο σας που έχετε για την, να ακούτε τη λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα παρουσιάσω πρώτα την εμπειρία μου και τα κίνητρα που με οδηγούν να ζητήσω την θέση αυτή και μετά θα προχωρήσω σε ορισμένα θέματα πολιτικής και οργάνωσης για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είμαι διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ιρλανδίας από το 2015. Πριν από αυτό ήμουν καθηγητής οικονομικών. Ε, ε, ε, σημαντικό έργο έρευνας για την παγκόσμια, τα παγκόσμια δημοσιονομικά και την ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση. Η εμπειρική φύση της έρευνάς μου με οδήγησε να συνεργαστώ με πολλούς οργανισμούς που ασκούν πολιτική από το 1990 και μετά. Μεταξύ αυτών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον ΟΟΣΑ, την Διεθνή Τράπεζα ε, ε, συμψηφισμών και άλλες. Το 2001 είχα την τιμή να λάβω γερμανική, το γερμανικό βραβείο Μπέρνασέ για ε, ιδιαίτερες συμβολές στα νομισματικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει κρίσιμο ρόλο στην διαχείριση των οικονομικών και της δημοσιονομικής παγκοσμιοποίησης το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτρέψει στις χώρες μέλη να ε, αποφεληθούν από τις τέσσερις ελευθερίες και ταυτόχρονα να παίξει ισχυρό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Η Νομισματική Ένωση ιδίω έχει τη δυνατότητα να είναι πολύ αποτελεσματικός μηχανισμός για τη διαχείριση της δημοσιονομικής παγκοσμιοποίησης. Έχοντας κοινό νόμισμα, οι χώρες μέλη είναι λιγότερο ευάλωτε σε εξωτερικά σοκ από ε, τις ε, συναλλαγματικές αναταράξεις και ταυτόχρονα αυτό αποτελεί και μια προστασία σε περιπτώσεις, σε περιόδους κρίσεων. Αποκλείοντας νομισματικούς κινδύνους εντός της Ευρωζώνης, η, Ευρωπα... η Ένωση επιτρέπει να γίνει βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών της. Η κρίση αποκάλυψε σημαντικές ανεπάρκειες στο αρχικό θεσμικό πλαίσιο. Ωστόσο, η θεμελιώδης λογική παραμένει ισχυρή οι μεταρρυθμίσεις που ήρθαν μετά την κρίση έχουν ενισχύσει την αθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, έστω και αν παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή πλατφόρμα για σταθερότητα και ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό έχει καθορίσει όλη μου την πορεία έω τώρα, μεταξύ αυτών και την μετάβασή μου στην Κεντρική Τράπεζα του 2015, καθώ και τώρα την πρόταση τη υποψηφιότητά μου για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να έρθω τώρα, αν ε, συμφωνείτε, σε ορισμένα θέματα πολιτική και οργάνωση. Η βασική πρωταρχική εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι να υλοποιήσει την σταθερότητα τιμών στην ζώνη ευρώ. Το επέτυχε αυτό μέχρι την κρίση. Ωστόσο, χρειάστηκε να λάβει και ορισμένα μη συμβατικά μέτρα. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει επιτρέψει να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, να διατηρηθεί ο πληθωρισμός στα κατάλληλα πλαίσια, να μειωθεί ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού και σύν χρόνο να υπάρξει μια σύγκληση προς τον κοινό στόχο. Είναι σημαντικό ότι η στρατηγική βασίζεται σε δεδομένα και επιτρέπει την προσαρμογή στις αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Από το 2015 συμμετέχω σε αυτές τις αποφάσεις και αυτό το μείγμα ποσοτικής ανάλυσης και ανάπτυξης των οικονομικών μοντέλων έχει επιτρέψει στο Governing Council να λαμβάνει αποφάσεις με αυστηρό τρόπο, βασισμένο απόλυτα σε δεδομένα και να κατανοεί σωστά, να κατανοούν σωστά μάλλον οι συμμετέχοντες στις αγορές. Η δε εμπειρία μου με επέτρεψε να συμβάλλω σημαντικά στη διαδικασία αυτή. Να έρθω τώρα <clears throat> στον ρόλο της Κεντρική τραπεζά, Τράπεζας για την διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας παίζει ρόλο και για το μετριασμό των κινδύνων, αλλά και για την διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις επεισοδίων αστάθειας. σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του κινδύνου, υπάρχει το Financial Stability Report που είναι πολύ σημαντικό. Οι δε μακροπροληπτικές αρμοδιότητες τις παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Υπάρχουν και δύο μηχανισμοί, μακροπροληπτικό φόρουμ και μακροπροληπτικό bulletin, που επιτρέπουν την παρακολούθηση των κινδύνων. Είναι επίση σημαντική η συνεργασία της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με άλλους θεσμικούς οργανισμούς για τον συντονισμό της μακροπρολητικής πολιτικής ολόκληρη την Ευρώπη. Έχω συμμετάσχει στις ε, υποθέσει αυτές ως σύμβουλος και ως πρώην ε, ε, επικεφαλής τη Συμβουλευτική Τεχνικής Επιτροπής. Έχω ηγηθεί επίση τριών συγκεκριμένων project, την πρόσφατη High Level Task Force για ασφαλή στοιχεία ενεργητικού και την έκθεση του 2016 για την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Η πορεία μου στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, η οποία επίσης ε, είναι η κεντρική εθνική μακροπροληπτική αρχή, μακροπροληπτική αρχή. Εκεί έχουμε χρησιμοποιήσει συστήματα προστασίας όπως ε, το SII. Επίσης, η μακρά μου επιστημονική καριέρα μου επιτρέπει να έχω ε, σημαντικά, σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό. Τώρα να έρθω ε, λίγο ε, στην εποπτεία. Ο ρόλος αυτός για μένα είναι πολύ σημαντικός, διότι εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή, σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Είναι σημαντικό το έργο εποπτείας να ξεχωριστεί από τις άλλες λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά να υπάρχουν βεβαίως και αναγκαίες διασυνδέσεις μέσω των αναγκαίων μηχανισμών. Κατά την άποψή μου, αυτά, αυτοί οι τομείς θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Και ο συνδυασμός μεταξύ SSM της Οδηγίας για την εποπτεία και το Resolution Board θα δούμε μια συνεχή εξέλιξη η οποία θα πρέπει να περιλάβει σύν το χρόνο και την σταδιακή εισαγωγή του συστήματος ε, εγγύησης καταθέσεων. Έχω άμεση εμπειρία στην εποπτεία των μέτρων αυτών τα τελευταία χρόνια ως μέλος της Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα πέραν από την Τραπεζική Ένωση θεωρώ ότι κεφαλαιακές, η Ένωση Κεφαλαιακών Αγορών είναι ένα σημαντικό θεμέλιο ακόμη για ένα πιο ισχυρό ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα. Και ιδίω για τις αγορές ε, αξιογράφων, όπου χρειάζεται αυτή η εποπτεία διαμεθοριακά. Επιτρέψτε μου να έρθω τώρα στις ε, δημοσιονομικές απαιτήσεις. Είναι προφανές ότι η σταθερότητα της Ευρωζώνης χρειάζεται συμμετοχή όλων των χωρών μελών για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Τελευταία, θα πρέπει μάλλον οι χώρες μέλη να ενισχύσουν τη δημοσιονομική τους σταθερότητα και με την εφαρμογή αντικυκλικών μηχανισμών να εξασφαλίσουν την ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης ότι δομικές πολιτικές θα ενισχύσουν την θέση των χωρών μελών και για την αντιμετώπιση κυκλικών σοκ. Αν σκεφτούμε τώρα τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, είναι σαφές ότι μηχανισμοί συνεργασίας των χωρών μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα εργαλεία για την αντιμετώπιση των ασυμμετρικών κραδασμών και μπορεί έτσι να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση σημαντικών κραδασμών όπως μια παγκόσμια ύφεση. Ο μηχανισμός σταθεροποίησης λοιπόν, η σταθεροποίηση μάλλον είναι σημαντικός στόχος και πρέπει να συνδέεται με πρωτοβουλίες για τη συνεργασία. Οι χώρες μέλη βέβαια θα αποφασίσουν για το μέλλον της δημοσιονομικής πολιτικής ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βέβαια βελτιώνεται εφόσον, ε, μάλλον διευκολύνεται εφόσον υπάρξει πρόοδο στου τομεί αυτού. Τέλο, να, να επανέλθω στην οργάνωση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου να είναι δεσμευμένα στην εξασφάλιση του ότι θα εργάζεται αποδοτικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τρόπο προοδευτικό και διαφανή, να είναι υπόλογη στους μετόχους της και να εξασφαλίζει τις ευέλτιστες συνθήκες εργασίας των μελών του προσωπικού της. Πρόσφατα λάβαμε βραβείο διαφάνειας από το transparency.com. Σωστό είναι να δημοσιεύονται όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, όπως πράττουμε δηλαδή. Επίσης είμαστε ηγέτης σε, στις προσπάθειες αυτές και δεσμευόμαστε και απέναντι στο προσωπικό μας για την παροχή κατάρτισης. Ελπίζω ότι θα μπορέσω όλα αυτά για την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Ε, ελπίζω ότι θα μπορέσω να μεταφέρω όλα αυτά εφόσον ε, διοριστώ στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έτσι ώστε να ενισχυθεί το κύρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Προ τα έξω και προ τα μέσα. Ελπίζω ότι με την συγκεκριτική μου αυτή τοποθέτηση θα συμφωνήσετε ότι θα είναι σημαντική η τοποθέτησή μου εκεί και ελπίζω πολύ να έχω την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λέιν για την πολύ, για την πολύ ενδιαφέρουσα αρχική σας παρουσίαση. Πρώτος ο κύριος Φέρβερ. Ευχαριστώ κύριε Λέιν, με μεγάλη χαρά σας βλέπω εδώ και ελπίζω, μια και είστε άλλωστε και ο μοναδικό υποψήφιο και σα έχουμε ήδη γνωρίσει, θα μπορέσουμε να οργανώσουμε μια ε, σωστή συνεργασία μεταξύ ημών και τη οικονομική επιτροπή. Θα ήθελα να μπω λίγο σε περισσότερη λεπτομέρεια στο ζήτημα πώ οι μηχανισμοί που έχει στη διάθεσή τη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιούνται πλήρω ή ποιου μηχανισμού βλέπετε, διότι υπάρχουν κάποιες σκιές ε, ήδη στην δραστηριότητα της ε, Ευρωζώνης, χωρών μελών τη Ευρωζώνης που ήδη έχουν μπει σε μια ύφεση ορισμένε εξ αυτών. Δεν βλέπουμε ε, τεράστια δυνατότητα ανάπτυξης. Βλέπουμε να διαμορφώνεται και ένας ακήρυκτος πόλεμος εμπορικού χαρακτήρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μηδενικά επιτόκια, με την ποσοτική χαλάρωση κλπ. Ποιους άλλους μηχανισμούς βλέπετε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και Μία προσωπική παρατήρηση για την πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για να εισπράξει αρνητικά επιτόκια. Εκπλήξει αυτό για μένα. Έχετε κάποια άποψη σχετικά. Διότι φαίνεται πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το θεωρεί αυτό ως το τελευταίο μέσον που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Θα ήθελα κάποια τοποθέτηση δική σας από αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. να ξεχωρίσω τις ερωτήσεις. Ένα είναι το πώς θα πρέπει να δούμε την απάντηση της Κεντρικής Τράπεζας στα αρνητικά νέα Βλέπουμε δύο πράγματα να προκύπτουν. Πρώτα απ' όλα ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παραμένει ε, ισχυρή ε, και πέφτει ενεργεία ιδίως στις αγορές όπου η ανεργία είναι χαμηλότερη από αλλού βλέπουμε να υπάρχει πίεση προς τα πάνω. Έχουμε λοιπόν την πεποίθηση ότι οι μηχανισμοί που θα επέτρεπαν να βελτιωθούν οι επιδόσεις στον πληθωρισμό προς στιγμήν ε, ισχύουν. Από την άλλη, από άλλους δείκτες είναι σαφές και από πολλές μελέτες προκύπτει ότι υπάρχει και μια λιλουχία από αρνητικές, ε, αρνητικά σοκ το τελευταίο διάστημα. Νομίζω λοιπόν λογικό είναι να πούμε ότι όλα αυτά βρίσκονται στην ε, περιοχή, στο χώρο της ανάγκης σχετικών προσαρμογών στις προβλέψεις. Δηλαδή θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες αναθεωρήσεις, κάποιες διορθώσεις, ε, χαμηλώνοντας τις αρχικές μας προσδοκίες κράτη-μέλη ε, ζήτησαν κάποια καθοδήγηση. Όταν, ας πούμε, τεπτόκια ε, ήταν ε, τάδε βασικά σημεία και βλέπουμε ότι σχετίζονται παρόλα αυτά και δεσμεύονται από την πραγματική οικονομία, έπρεπε να αλλάξουν. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο οι συντελεστέ σήμερα, αλλά και για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Υπάρχει συσχετισμός διότι τα θεμέλια για τα μελλοντικά επιτόκια είναι το τι θα κάνουν οι αγορές ε, όχι μόνο φέτο, αλλά και του χρόνου και του παραχρόνου και ούτω καθεξή. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντε και άλλοι παράγοντε που ενεργοποιούνται, αλλά αυτό είναι ένα μέλο του μεγάλου πολιτικού πακέτου σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση αυτή τη στιγμή. Ότι προ στιγμή τα στοιχεία δείχνουν από το περασμένο καλοκαίρι ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στα επιτόκια μετά το καλοκαίρι. Και μετά αυτό θα, εξελιχθεί και από θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το, ε, με το πώς βλέπουμε τις προβλέψεις. Αφού η αγορά, εάν δούμε τι θα γίνει με τα επιτόκια στο μέλλον, η αγορά προσδοκά να γίνει διόρθωση προς τα κάτω, αλλά με χαμηλότερο, με αργότερο, βραδύτερο ρυθμό από το προηγουμένω. Οπότε μακροπρόθεσμα η στρατηγική μα πρέπει αυτό να κοιτάξει να αντιμετωπίσει. Τώρα, αν έχουμε μεγάλο σοκ, ε, αρνητικότερο πλήγμα από ό,τι υπολογίζουμε, ο πληθωρισμό όχι απλώ θα επιβραδυνθεί, αλλά θα αντιστραφεί. Η τωρινή μα στρατηγική έχει δείξει ότι πάνω απ' όλα θέλουμε να πετύχουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους. Και παρόλο που έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία, Δεν νομίζω ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει ξεπεράσει όλα τα όρια και έχει αξιοποιήσει όλες τις ε, δυνατότητες. Και καλό θα ήταν να μην είμαστε και πάρα πολύ συγκεκριμένοι και ακριβεί στο τι συνδυασμό εργαλείων θα χρησιμοποιήσουμε. Ε, είναι πολλά τα πρακτικά εδώ. Μακροπρόθεσμα μιλήσατε και για τι γενικέ επιπτώσει στη ρευστότητα. Αυτό δεν το βλέπω ως κάτι που θα προκύψει άμεσα, αλλά αν κοιτάξει κανείς σε έναν ορίζοντα όχι δεκαετίας μόνο, αλλά αρκετών δεκαετιών, υπάρχει ένα θέμα. Ποιο ήταν ο ρόλος των μετρητών της ρευστότητας στο μέλλον. Μήπως γίνουν κυρίως ηλεκτρονικά και είναι λιγότερο και αυτά που έχει στο, στη διάθεση του το κράτος και, και από τους φόρους. ηλεκτρονικό χρήμα τα κυκλοφορεί και ίσως τεχνικός να είναι δυνατόν να έχουμε και αρνητικά επιτόκια ή φόρους σε αντιστοιχίες ρευστότητας. Κάποιοι θα σας πούν ότι αυτό είναι ίσως το μέλλον, αλλά μεσοπρόθεσμα δεν ξέρω αν θα συμβεί. Δεν βλέπω τα μετρητά να εξαφανίζονται σύντομα. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε, αλλά Σίγουρα πρέπει να γίνει κάποια έρευνα, να δούμε τι θα γίνει στο απότερο μέλλον, αλλά δεν είναι προ στιγμή κάτι που θα μα αποσχολήσει αμέσω, πιστεύω. Ευχαριστούμε, περιμένεις; Μερές. Μία ερώτηση Θα ήθελα μία απάντηση, μία ερώτηση ολικής αχνίας να σας κάνω. Με ναι ή όχι θα ήθελα την απάντηση. Ε, ναι ή όχι, πείτε μου. Τι σημασία αποδίδεται, μάλλον αποδίδεται σημασία στο νομισματικό διάλογο μεταξύ ΕΚΤ και Ευρωκοινοβουλίου. Ναι. Ωραία. Στη γραπτή ερώτηση που σας απέστειλε, η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ρωτάει αν θα δεχτείτε το διορισμό στο εκτελεστικό ε, συμβουλίο του ΣΕΚΤΕ, αν καταψηφίσετε την υποψηφιότητά σας ε, το Κοινοβούλιο. Και λέτε ότι χαίρομαι που με πρότεινε η κυβέρνησή μου και με δέχτηκε το Συμβούλιο ελπίζοντας ότι και το Κοινοβούλιο θα ε, υπερψηφίσει την ε, άποψη του Συμβουλίου. Θεωρείτε ότι είναι μια ορθή απάντηση αυτή? Ε, κοιτάξτε, ε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι σαφές ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ στη διαδικασία διορισμών, που είναι διαφορετικό πράγμα από το νομισματικό διάλογο. Νομίζω λοιπόν ότι θα ακολουθήσω τους κανόνες, όπως έχουν σχεδιαστεί από άλλους. Θέλω όμως, επειδή παρακολουθώ το νομισματικό διάλογο ακόμα και τώρα, και επειδή είμαι και ακαδημαϊκός, ο νομισματικός διάλογος είναι ένας πολύ αποδοτικό τρόπος να ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ενημερωτικά και συμβουλευτικά ε, δελτία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, οι δημοσιογράφοι θέτουν ερωτήσεις. Οπότε είναι σαφώς πολύ πρόσφορος ο διάλογος εδώ. Ε, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διάλογος. Είναι κέρια σημασία, ήδη έχει μεγάλη σημασία και αυτό φαντάζομαι θα ισχύει και στο μέλλον. Τώρα για τη διαδικασία διορισμού θα ήταν ανάρμοστο να κάνω περαιτέρω σχόλια. Δεν μπορώ εγώ να καθαρίσω τη διαδικασία διορισμού. Αποδίδεται σημασία στον νομισματικό διάλογο. Θεωρείται ότι ακαδημαϊκό είναι πολύ καλό, ένα επιπλέον εργαλείο. αλλά δεν θα σας πείραζε να είσαστε μέλος της Κεντρικής Τράπεζας κατά αντίθετα με την άποψη του Κοινοβουλίου. Εμεί εδώ δεν είμαστε όμω ακαδημαϊκοί, δεν είμαστε πανεπιστημιακοί, δεν είμαστε εδώ απλώ για να ομορφύνουμε τη συζήτηση για την ε, νομισματική πολιτική. Εάν υπάρχει στρέβλωση στο κάτω δικαίου που τη θεωρούμε ε, μη λογική, ε, όχι. Εάν συγκρίνεται την κατάσταση τη Κεντρική Τράπεζα με τη ΦΕΔ, εάν το Κογκρέσο, αν το ας πούμε, είχε αντιταχθεί στην, ε, στο, σε κάποιο διορισμό, δεν θα γινότανε. Λέτε λοιπόν ότι ο νομισματικό διάλογο είναι χρήσιμο, αλλά εμεί καλούμε το Συμβούλιο να λάβει υπόψη και την άποψη του Κοινοβουλίου. Αυτό μα ενδιαφέρει να συμβεί. So, I think uh, for anyone going for... Όποιο πηγαίνει για το εκτελεστικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο δηλαδή. Καλό θα ήταν να έχετε την υποστήριξη και του Ευρωκοινοβουλίου. Ούτω ή άλλως. Αλλά δεν είμαστε πολιτικοί. Και νομίζω ότι το πώς έχει καταρτιστεί η διαδικασία διορισμού είναι κάτι που το πολιτικό σύστημα πρέπει να το αποφασίσει, όχι εμεί. Προβλέπονται οι ευθύνε από το ίδιο το σύστημα τη διαδικασία. Δεν μπορώ εγώ να τι αποφασίσω τι ευθύνε αυτέ. Βεβαίω στι ΗΠΑ το, το σύστημα είναι διαφορετικό. Χρειάζεται η έγκριση από το Κογκρέσο. Αλλά για μένα είναι σαφώ πολύ σημαντική άποψη του Ευρωκοινοβουλίου. Και βεβαίω θα τη λάβει υπόψη και το Συμβούλιο αυτή την άποψη. Το ότι έχετε συμβουλευτικό ρόλο εδώ, ε, σαφώς σας κάνει βαρύνουσα σημασία για την τελική απόφαση. Ευχαριστούμε. Πακέτα από το ECR τώρα. Ευχαριστώ. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Εάν η Ευρωζώνη μπει σε ύφεση πριν προλάβει να αυξήσει τα επιτόκια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εσείς μπορείτε να φανταστείτε αρνητικά επιτόκια και πώς τι επιπτώσεις θα έχουν στην διάθεση ρευστού. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, Πιστεύετε ότι η νομισματική πολιτική μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση και πιστεύετε ότι είναι στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ. Απάντηση. Όπως γνωρίζετε, ξέρουμε ότι δεν βρισκόμαστε σε αρνητικό επίπεδο και οποιαδήποτε εκτίμηση συνδυασμού ε, προγραμμάτων αγοράς ομολόγων ή αλλαγή στα επιτόκια. Είναι ένας συνδυασμό. έπειτα υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές. Όπως είπα πριν, όταν έχουμε να κάνουμε με μία υποθήκη, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο τα σημερινά επιτόκια, αλλά ποια θα είναι η εξέλιξή του στο μέλλον επίσης. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να ξέρουμε όχι μόνο το τι συμβαίνει σήμερα, αλλά και ποιες είναι οι προβλέψεις για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν συνδυάζει όλα αυτά τα εργαλεία με αρνητικά επιτόκια. Αν πάνε πολύ στο μείον, δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν και πρέπει φυσικά να γίνει η εκτίμηση. Όσον αφορά τη ρευστότητα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, εννοείται ότι έχει το 0%, αν όμως πάμε πιο αρνητικό, ο κόσμος μπορεί να φοβηθεί για το ρευστό που κρατάει. Αλλά αυτός ο κίνδυνος είναι κάτι που μπορούμε να διαχειριστούμε με διάφορους τρόπους. Για το μέλλον αν έχουμε λιγότερο ρευστό θα είναι λιγότερο προβληματικό. Όλα όμως έχουν να κάνουν με τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Αν οι συνθήκες είναι τέτοιες όπου έχουμε αδύναμη οικονομική ε, απόδοση, τότε πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί είναι ζωτική σημασία. Και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ακριβώς να είναι σαφής ότι σέβεται τους μεσοπρόθεσμους στόχους. Και αυτό ακριβώς κάνει με τα μέτρα που παίρνει. Τώρα για το μακροπρόθεσμο. Τι θα οδηγήσει σε ευημερία. Είναι η παραγωγικότητα, είναι οι επενδύσεις, είναι η εκπαίδευση, είναι καλοί θεσμοί. Ό,τι τα καταστρέφει αυτά οδηγεί αστάθεια. Μια καλή πάντως πολιτική σημαίνει ότι και άλλες πολιτικές να πάρουν την σημασία που τους πρέπει. Γιατί αποτελούν παράγοντα σταθερότητας πάντα. Ευχαριστούμε, Λέω Πρόεδρος Καρβέ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βλακωνικά, κύριε Δικητά της Ιρλανδικής Κεντρικής Τράπεζας. Ξέρουμε όλοι ότι είσαστε καλά προετοιμασμένος για να λάβετε αυτά τα καθήκοντα και ξέρετε πολύ καλά από στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας ακαδημαϊκά. Η ερώτησή μου είναι εξής. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης, εσείς τι πιστεύετε ότι μείωσε την, ε, τον ευάλωτο χαρακτήρα του ευρώ γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα λιγότερο μέχρι την επόμενη κρίση. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν ελήφθησαν αρκετά μέτρα για να γίνει λιγότερο ευάλωτο το ευρώ. Εσείς τι πιστεύετε επίση για τα μη συμβατικά μέτρα που εφαρμόστηκαν. Ε, κατά σύμπτωση, πρόσφατα έχουμε μια μελέτη που λέει ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις από την έξοδο από την κρίση. Πρόκειται για ένα Ολλανδικό Ινστιτούτο, έτσι να το πούμε και αυτό έχει και αυτό την σημασία του. Εσείς τι λέτε. Τρίτον, σας άκουσα και την προηγούμενη φορά που μιλούσατε για ε, το EBCC και για το πόσο το ενίο νόμισμα στηρίζει το όργανο αυτό. Τι πιστεύει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι θα μπορούσε να κάνει για να αντιμετωπίσει το κοινωνικό dumping που στη δικιά σας χώρα από την οποία θα φύγετε για να πάτε στην Φραγκφούρτη. Το έχει κάνει σημαία και παντιέρα, το κοινωνικό dumping. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά το θέμα της αρχιτεκτονικής, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι έχουν γίνει πολλά δημιουργήθηκαν οι εποπτικοί μηχανισμοί, ε, δημιουργήθηκε ο μηχανισμός ε, εξυγίανσης, δημιουργήθηκε ο ESM. Όλοι αυτοί οι παράγοντες προσφέρουν περισσότερη σταθερότητα σε περίπτωση επόμενης κρίσης. Δύο παράγοντες υπογραμμίζω. Πρώτον, να είμαστε σίγουροι ότι οι χρηματοπιστωτικές πολιτικές είναι καλές. Γιατί σίγουρα έχει γίνει πολύ πρόοδος. Αλλά ακόμα και τώρα το γεγονός ε, της ε, δημοσιονομικής πειθαρχίας Σήμερα η Ευρώπη είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει προβλήματα από ό,τι ήταν πριν από 5-6 χρόνια. Επίσης, φυσικά υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για τα κοινά ε, ε δημοσιονομικά. Όμως αυτό που έχουμε σήμερα είναι μια Ευρώπη που έχει λιγότερες ανισορροπίες από ό,τι κατά το παρελθόν, δεν βρίσκεται στην κατάσταση που βρισκόταν σε αρχές του 2000 της νέας χιλιετίας, έχουμε λιγότερα ελλείμματα, χρέη κτλ. Η Ευρώπη δηλαδή σήμερα δεν είναι σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση. Σίγουρα είναι σημαντικό να συνεχίσει η πρόοδος και όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις τράπεζες, φυσικά και πρέπει να συνεχίσουμε. Και είναι σημαντικό τελικά να καταλήξουμε να έχουμε ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Πάντως υπογραμμίζω ότι σε σύγκριση με το που βρισκόμασταν πριν από χρόνια έχει επιτευχθεί τεράστια πρόεδρος. Τώρα, πρόοδος. Τώρα για τις μη συμβατικέ ε, πολιτικές. Είμαστε θετικοί. Το γεγονός ότι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο από το καλοκαίρι του 2014 και με την αγορά ενεργητικών στοιχείων, με την έγκριση των τεσσάρων κατευθυντηρίων γραμμών, όλα αυτά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και έχουμε πολύ καλύτερε συνθήκε στην αγορά σήμερα από ό,τι είχαμε πριν από πέντε χρόνια στην Ευρώπη. Και αυτό φαίνεται και από την πιστοτική ικανότητα και κατάσταση, από την ανάκαμψη παντού στην Ευρώπη. Οπότε, πιστεύω ότι δεν επιτυχεί τα μέτρα. Αυτά όσον αφορά το μέλλον, για εδώ, Αμερική και τα λοιπά, η εξωτερικεύση σίγουρα έχει, χρειάζεται κάποια εξισορρόπηση. Και τώρα για τη σημασία που έχει η συνέχεια στην Ευρώπη και η ενιαία αντιμετώπιση. Όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα, η λύση δεν είναι η αμοιβεποίηση. Και εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε με τις πολιτικές αποφάσεις. Γιατί αν υπάρχει τέτοια αμοιβεποίηση, ποια θα είναι. Τι δυνατότητες υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Θέλουμε να έχουμε κοινά ομόλογα χωρίς ε, αμοιβεποίηση. Μπορεί κάτι τέτοιο να προσφέρει πρόοδο. Τώρα, το τελευταίο, ρωτάτε για τον εταιρικό φόρο ουσιαστικά. Και πάλι στη γραπτή μου απάντηση το έχω πει ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και ευρωπαϊκό ζήτημα. Ότι έχει να κάνει με τις σχέσεις των χωρών μεταξύ τους και με τις επιχειρήσεις. Η κάθε χώρα έχει διαφορετική κατάσταση, αλλά απαιτείται μια ευρωπαϊκή και μια παγκόσμια ε, απάντηση που να ισχύει παντού. Αλλά το πολιτικό σύστημα θα την πάρει αυτή την απόφαση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ορτασούν. Ευχαριστώ κύριε Λέιν παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον την τελευταία παράδοση στο Galway, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας και σε σχέση με τις ε, κλιματικές αλλαγές. Εκεί στη διάλεξή σα είπατε ότι οι κεντρικέ τράπεζε έχουν ευθύνη να βεβαιωθούν ότι οι θετικέ πατεριότητε με τι κλιματικέ αλλαγέ ε, συνδυάζονται στο με το οικονομικό σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σα για το πώ η ΕΚΤ σκοπεύει να συνδυάσει του στόχου τη στι ευθύνε που δημιουργεί η Συμφωνία των Παρισίων ε, για τι κλιματικέ αλλαγέ. Υπάρχουν ανησυχίε για τα προγράμματα αγορών για τα περιουσιακά στοιχεία. Τα ενεργητικών στοιχείων. Και πώς θα κάνουμε κάτι για την αγορά των, του, των στοιχείων ενεργητικού, ε, των περισσιακών στοιχείων, ε, προσπαθώντας να το συνδυάσουμε με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για, την ε, για το ενδιαφέρον σας για τη διάλεξή μου. Οι κλιματικές αλλαγές ε, θα γίνουν προτεραιότητα και για την ΕΚΤ, καθώς θα γίνει και πολλά, ε, πολλούς κλάδους σχεδιασμού πολιτικής. Η απαλλαγή της οικονομίας από τον άνθρακα, ας πούμε, είναι σημαντικό. Για, την, ε, για το συνθισμό πολιτικών ε, είναι μία λύση. Αλλά εκεί που η οικονομική σταθερότητα αρχίζει δεν ε, πηγαίνει έκτη. Η οικονομική αστάθεια δηλαδή από στοιχεία του ενεργητικού που έχουν σχέση με τον άνθρακα, εκεί η ΕΚΤ θα πρέπει να αναλάβει μακροπροληπτικές ευθύνες. Χρειάζεται γίνονται δοκιμές ε, αντοχής, ανθεκτικότητας μάλλον, η δημοσιοποίηση των φορολογικών ε, στοιχείων, του φορολογικού αρχιτεκτονήματος και το τι γίνεται με τον άνθρακα. Οι επόπτες θα έχουν πολλή δουλειά σε σχέση με την καθοδήγηση που θα έχουν να δώσουν στους τράπεζες, την αξιόλογηση κινδύνων και το καθεξής. Ως προς την ε, πολυπολιτική, το συνδυασμό πολιτικών δηλαδή, δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, εάν τα σοκ, οι τρεγμοί έχουν σχέση με την διακύμαξη που βλέπουμε. Δεδομένου του τι συμβαίνει τώρα με τις διακοπές στην παραγωγή που έχουν να κάνουν με το ότι το καλοκαίρι είναι πολύ θερμό, ο χειμώνα πολύ ψυχρό ή υγρός και ούτω καθεξής. Αυτά πρέπει να μας κάνουν να μελετήσουμε πολύ καλύτερα τις υλικέ και οικονομικές συνέπειες των αλλαγών στο κλίμα, των διαφορετικών κύκλων που βλέπουμε. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή των ε, συνδυασμένων πολιτικών, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει μια τελική παρατήρηση, να βγάλει ένα τελικό συμπέρασμα. Πολλά γίνονται και βρίσκονται σε εξέλιξη. Βλέποντας ότι έχει προκύψει ως τώρα σε γραπτό κείμενο, σήμερα ο συνδυασμός αυτός πολιτικής δεν έχει γίνει κάτι το παγιωμένο, το καθ αφιερωμένο. Ε, τα πράσινα ομόλογα πούμε, δεν έχουν προχωρήσει ακόμη και αν υπάρξει μια προτίμηση για την ε, χαμηλή κατανάλωση άνθρακα με ένα πρόγραμμα ομολόγων λόγω χάρη στο ε, μέλλον. Θα είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώ θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Για να είμαι ειλικρινή, λοιπόν προ στιγμή το ζήτημα γίνεται δευτερεύον σε σχέση με την οικονομική σταθερότητα και την εποπτεία. Έρχεται λίγο δεύτερο. Αλλά θα τα δούμε στο μέλλον. Ο κύριος Κερέικ ε, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία πριν από λίγους μήνες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε το βλέμμα στραμμένο και προς το μέλλον. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω μιλητές από τις άλλες ομάδες. Κάτσε τώρα ο κύριος Λάνιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν επιθυμώ καθόλου να αμφισβητήσω τα προσόντα σας. Η γραπτή σας απάντηση για την, ε, μάλλον η πρότασή σας να απαντήσει γραπτό στην κυρία ε, Μπερές και εκεί συμφωνώ. Αλλά τούτη εδώ την τελευταία σας άρνηση να απαντήσετε δεν μου φαίνεται σωστή. Θεωρώ ότι ένα μέλος του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επιμένει ότι θα είναι ανεξάρτητο όταν θα αναλάβει τα καθήκοντά του, θα πρέπει να αποδεχτεί τις δημοκρατικές δομές. Ούτε μπορώ να φανταστώ ότι ο μελλοντικό πρόεδρος του, ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Συμβουλίου δηλαδή, ε, θα μπορούσε να αντιταχθεί σε μια αρνητική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί κάτι τέτοιο πιστεύω ότι στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία θα προχωρήσουμε σε διοργανική συμφωνία με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Όπως προ 15 ετία είχαμε κάνει ήδη με τον ε, τότε πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μπαρόσο, ο οποίος πρώτη εκλογής του είχε δηλώσει ότι ναι, κάθε επίτροπος ο οποίος ε, θα λάβει με ενισχυμένη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνητική ψήφο θα πρέπει να παραιτηθεί. Θεωρώ ότι για να προχωρήσετε να καταλάβετε θέση στο εκτελεστικό συμβούλιο τη Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να έχετε θετική ψήφο του Κοινοβουλίου και όχι να λέτε κατά βάση δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ τα άλλα θεσμικά όργανα με πρότειναν και ό,τι και να γίνει εγώ οπωσδήποτε θα, τοποθε, θα διοριστώ. Αρχικά δεν είχα καταλάβει το ιστορικό της ερωτήσεως της κυρίας Μπερές, αλλά σας παρακαλώ τώρα να τοποθετηθείτε και μάλιστα ξεκάθαρα. Just the point, because of course you... Ευχαριστώ. Ήταν πολύ άμεση η ερώτησή σα στον κύριο Λέιν. Αλλά από θεσμική σκοπιά, ενώ έχω κατανόηση για αυτά που λέτε, ο συνομιλητής εδώ είναι το Συμβούλιο. Έχουμε σύσταση του ΕΚΟΦΗΝ και σύσταση του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει. Δεν είναι πρόβλημα ατόμου, είναι πρόβλημα ε, βέβαια στι συνθήκε τα πράγματα λέγονται διαφορετικά. Έχουμε αυτό το μικρό πρόβλημα. Ότι οι συνθήκε δεν είναι δεσμευτικέ, άλλω ε, δεν θα ήταν σύμφωνη γνώμη. Αλλά πρέπει να απευθυνθούμε στο Συμβούλιο και να του πούμε πώ πολιτικώ αποτιμάται τη δική μα την τοποθέτηση. Ιδίω αν πάμε στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Αυτό για την ερώτησή σα. Εγώ νομίζω ότι η απάντηση δεν έχει να κάνει με τα θεσμικά που αφορούν εμά, μεταξύ μα. Ε, κοιτάξτε, θα διαφωνήσω εάν νομίζετε ότι δεν με νοιάζει. Και αν νομίζετε ότι την άποψή σας την έχω, ε, της δίνω μικρή σημασία. Ελπίζω πάντως να πάρω έγκριση και από εσά, γιατί στη διαδικασία έγκρισης, στην τελική απόφαση την έχει το Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι αδιάφορο ως προς την άποψή σας. Ε, κάθε άλλο. Αλλά δεν είναι δική μου η θέση να λάβω αποφάσεις για το πώ γίνεται ο διορισμό. Τα άλλα θεσμικά όργανα πρέπει να αποφασίσουν. Όχι υποψήφιο. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Ευχαριστούμε για αυτή την τόσο ωραία ανταλλαγή απόψεων και ελπίζουμε ότι τελική άποψή μας θα είναι και θετική. Ευχαριστούμε.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 So we move to point 11. I would like... Uh, Σημείο 11. Να καλωσορίσω τον κύριο Ζωζέ Μανουέλ Κάμπα. Όπως τα γνωρίζετε, επελεγεί από το Συμβούλιο Εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ως πρόεδρος τους, και αν επιβεβαιωθεί θα καλύψει τη θέση που προέκυψε από την παρέτηση του κυρίου Αντρέα Ενρία στις αρχές της χρονιάς. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ε, κοινοποίησε στο Ευρωκοινοβούλιο στις 19 Φεβρουαρίου την απόφασή της. Ο κύριος Κάμπα επελέγει από ένα κατάλογο υποψηφίων από την ε, Επιτροπή Επιλογής ε, της EBA. και θα έχουμε μια ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Κάμπα. Και τώρα βάσει των όσων ορίζουν οι κανόνες έχουμε αυτή τη διαδικασία που είναι κάπως ιδιότυπη του να δούμε αν θα προβάλλουμε κάποια μομφή για αντίρρηση ή όχι. Είναι πρόεδρος της CBA, ο Κάμπα. Είναι μια σημαντική λοιπόν στιγμή για να ε, αναδείξουμε ανάγλυφα την ε, ε, υποχρέωση λογοδοσίας της διοίκησης και διεύθυνσης της CBA προς το Κοινοβούλιο. Έχετε λάβει το βιογραφικό του κυρίου Κάμπα. Καλώς ορίσατε. Συγχαρητήρια για την ε, επιλογή σας από τους επόπτες. Σας δίνω το λόγο για μια αρχική εισήγηση και μετά θα κάνετε ε, διάλογο με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας μέλη της Επιτροπής. Για μένα είναι χαρά και τιμή μου να είμαι σήμερα μαζί σας. Μου ζητήσατε να κάνω μια σύντομη εισήγηση για να υποστηρίξω τον διορισμό μου ως Προέδρου της EBA, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Με ακούτε? Θα έχετε το λόγο πολύ σύντομα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι παρόλα όσα συνέβησαν, ο ρόλο τη είναι ουσιαστική σημασία και σήμερα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή μα λειτουργία για να υπάρχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο για όλο τον τραπεζικό κλάδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει διαφανή και ε, λειτουργική ε, αγορά για του Ευρωπαίου καταναλωτέ και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η εντολή μα είναι επίκαιρη και σήμερα και θα πρέπει να μα καθοδηγήσει την ερχόμενη πενταετία. Η εντολή αφορά τρεις βασικές δραστηριότητε της ε, EBA, το ενιαίο τραπεζικό χειρίδιο για τις τραπεζικές δραστηριότητε, τις πρακτικές λογοδοσίες και την ενερμονισμένη εφαρμογή των κανονών διάσωσης, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας ε, και γενικότερα την εξυγένση του τραπεζικού κλάδου με πολλά εργαλεία, τον εντοπισμό της βαλωτότητα, της, ε, του, κατά πόσων οι τράπεζες είναι βάλωτες, Ε, και τον ε, τεστ αντοχής. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές και στο μέλλον για να τις αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. οι τραπεζι, ο τραπεζικός κλάδος, οι τράπεζες γενικότερα θα αλλάξουν πολύ τα ερχόμενα χρόνια. τεχνολογία και οι πετήσεις των πελατών επηρεάζουν τον κλάδο. Επίση, η δημιουργία τη ενιαία αγορά και η Τραπεζική Ένωση σίγουρα θα προκαλέσουν και άλλε διαθετικέ αλλαγέ. Η ABA είναι σε θέση να αναλάβει το ρόλο τη εδώ βασιζόμενη στην εμπειρία τη. Για την τελευταία δεκαετία έχει συγκεντρώσει πολλή τεχνογνωσία για τη λειτουργία του τραπεζικού κλάδου και αυτή η τεχνογνωσία είναι μοναδική και θα συνεχίσει να διωγγώνεται και στο μέλλον. Η EBA θα μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση της δράσης μας στην μεταβατική περίοδο με πέντε βασικά θέματα που ήδη αντιμετωπίζουμε εν μέρη. Πρώτα απ' όλα να αναπτύξουμε τους κανόνες. Να υπάρχει μια εύρυθμα λειτουργώσα ε, εσωτερική αγορά κλίμα προστασία των καταναλωτών. Δεύτερο, η προσαρμογή των τραπεζών και του τραπεζικού πλαισίου στι νέε ανάγκε και τι τεχνολογικέ εξελίξει. Η EBA ήδη έχει αρχίσει τη δουλειά τη σχετικά. Έπειτα, σύγκληση των καλύτερων ε, διαδικασιών εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερα, ε, πληροφορία και ενημέρωση για, το, για την κατάσταση του κλάδου και το πώς λειτουργεί όλος ο κλάδος για την ε, καταγραφή των κινδύνων και τα χαρακτηριστικά των τραπεζών. καθώς και το ποιες είναι οι καλύτερες ρυθμιστικές και εποπτικές πρακτικές. Η EBA θα έχει ενεργότερο ρόλο στο να φέρει την γνώση αυτή ε, στο φως για τους επιτρόπους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορέσουν αυτές οι λειτουργίες να καταπτυχθούν σωστά. Επίσης, βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ε, της ανάγκης για τον Brexit, που είναι ένα μείζονο σημασίας γεγονός, και μετά να έχουμε μια καλά διαρθρωμένη συνεργασία με τρίτες χώρες για τα ειδικά καθεστώτα και την φορολογική μας συνεργασία. Τέλος, να τονίσω ότι η EBA θα πρέπει να ελάβει το ρόλο της, ε, έχοντας υπόψη το τι είναι κατάλληλο για ποιον, πότε και γιατί. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάγνωση για τις θεσμικές δραστηριότητε που διθετώνται και τα άλλα ε, εμπλεκόμενα ζητήματα. Η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνεται. Κάποιοι κανόνε όπω προστασία των καταναλωτών, η δημοσιοοικονομική σταθερότητα, η πρόσβαση τη υπηρεσια και ανταγωνισμό, η προστασία τη ενή αγορά πρέπει να είναι οριζόντιο χαρακτήρα. Άλλα εργαλεία, η υποχρέωση υποβολή εκθέσεων λόγω χάρη, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αναλογικώ μόνον ώστε οι στόχοι να επιδιώκονται και να επιτυγχάνονται χωρίς να επηρεάζουμε ε, όσους λειτουργούν στον κλάδο, ιδίω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι φιλόδοξη η ατζέντα μας, αλλά για τα ερχόμενα πέντε χρόνια στην EBA ελπίζω ότι θα μπορέσω να συνεισφέρω στην επίτευξη των στόχων μας. Let me thank you again for having me here. Σας ευχαριστώ ξανά που με καλέσατε σήμερα και μου δώσετε την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο. Ε, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, για την ε, αρχική σας τοποθέτηση. Πρώτος λαμβάνει το λόγο ο κύριος Μπάρκος Φέρβερ. Ευχαριστώ κύριε Κάμπα. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω γερμανικά και μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μετάφραση. Ελπίζω ότι ε, κατανοείτε τι λέω τώρα. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτο, Έχουμε τώρα οδηγία και κανονισμό για τα ίδια κεφάλαια και θα ψηφίσουμε σήμερα για την έκβαση του τριμερούς διαλόγου. Έρθω, ε, θα ήθελα να, ε, να, ρωτήσω για την αναλογικότητα, για το γραφειοκρατικό βάρος των ε, μικρών κυρίως πιστοτικών ιδρυμάτων, το οποίο καλείται να μειωθεί κατά 10%. Πώς το βλέπετε. Δεύτερο, η αρχή της τραπεζικής εποπτείας προχωρεί, έχει συμφωνήσει μάλλον για την ε, θέσπιση της Βασιλείας 3. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Για τη δέσμη μέτρων της Βασιλείας 3 έχετε άποψη, θα πρέπει να την δεχθούμε 100% όσο έχει ή θα πρέπει να επιφέρουμε κατά την άποψή σας κάποιες αλλαγές. Αυτές είναι οι δυο μου ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά την αλογικότητα. Ίσως ακούσατε και από την ομιλία μου ότι θα πρέπει να είναι μια θεμελιώδης αρχή αν κατάλαβα καλά από την ερώτησή σας, αυτό στοχεύει κυρίως στην ε, διοικητική επιβάρυνση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη λοιπόν η θεμελιώδης αυτή η αρχή, ώστε να υπάρξει η σωστή αναλογικότητα ε, στην νομοθεσία, ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο που θα επιλεχθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή είναι η απόφαση που έχει ληφθεί στο παρελθόν, έχει εγκρίνει τις απαιτήσει της Βασιλείας για όλα τα τραπεζικά ιδρύματα. Και αυτή υπήρξε απόφαση Και νομίζω ότι τώρα πρέπει να συνεχίσουμε στην πορεία αυτή. Νομίζω ότι οι εξελίξεις δείχνουν άλλωστε προς την κατεύθυνση αυτή και αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει και τα επιχειρηματικά μοντέλα και την διαμόρφωση, τη διάρθρωση των τραπεζών στην Ευρώπη. Χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. για να υπάρχει δυνατότητα μέσω των διαδικασιών εξηγένσης να μην επιβαρυνθεί η δημοσιονομική σταθερότητα ούτε οι καταθέσεις των αποταμιευτών. Όχι μόνο λοιπόν η αναλογικότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη, στη κοινωνική επιβάρυνση αλλά και σε όλα τα σχετικά μέτρα. Ο κύριος Φέρμπερ, απαντήσατε πράγματι ταχύτητα, ε, πολύ σύντομα ακόμη. Ήσασταν και chief lobbyist της Banco Santander, μιας μεγάλης τράπεζας δηλαδή. Θεωρείτε ότι είναι ε, διασφαλισμένη η ανεξαρτησία σας στο μέλλον, εφόσον καταλάβετε τη θέση που επιθυμείτε. Όπως το μετέφρασαν την ε, ερώτησή σας μπορώ να απαντήσω απλώς ναι. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συλλέξει ε, σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Τα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια βεβαίως συνέβαλαν στην επαγγελματική μου ανέλυξη, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Έχω εμπειρία την οποία θα μεταφέρω στις εργασίες μου στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. θεωρώ ότι η εμπειρία αυτή αυξάνει την δυνατότητα κατανόησής μου των διαφόρων συσχετισμών, των μηχανισμών και των μέτρων που θα απαιτηθούν για να υπάρξει μια σωστή λειτουργία του τραπεζικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Αυτά, ε, λόγω του ιστορικού μου ε, και στο Πανεπιστήμιο, αλλά και ως δημόσιος λειτουργός. Και νομίζω ότι η εμπειρία μου αυτή μου προσφέρει ε, και μια ε, μοναδική οπτική για το πώς ε, εξετάζω τον κλάδο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μπερές. Και εγώ θέλω να συνεχίσω μετά από την τελευταία ερώτηση. Από το 2014 είσαστε στην τράπεζα αυτή Ταντερ, και ασχολείστε με τα ρυθμιστικά ζητήματα, αυτά που έχουν να κάνουν με την τραπεζική αρχή. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι too close to speak όταν οι υπόπτες δηλαδή έχουν τόσο στενή σχέση με μια τράπεζα ε, πώς μπορείτε να διασφαλίσετε το ρόλο σας. Οπότε αυτή είναι η ερώτησή Πώς βλέπετε εσείς τις επαφές με την τράπεζα του Σανταντέρ τη στιγμή που θα σας ζητήσουν αυτή την επαφή. Δεύτερον, για την νομοποίηση παράνομου χρήματος. Γνωρίζετε ότι σήμερα γίνεται μια αναθεώρηση στις εποπτικές ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου η EBA να αποτελέσει μια πλατφόρμα. Εσείς πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτή, την ευρωπαϊκή μάχη δηλαδή για την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομου χρήματος και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συνεργασία του εποπτικού σκέλους του FIUs. Νομίζετε δηλαδή ότι η EBA θα φτάνει για να ασχοληθεί με ολόκληρα τα θέματα του συντονισμού του FIUs ή βλέπετε κάποιες άλλες εξελίξεις ως αναγκαίες εσείς. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για τη σχέση μου με την τράπεζα Σανταντέρ, αν σας κατάλαβα καλά, λέτε πώς θα διαχειριστώ την σχέση μου μαζί τους εφ' εξής. Μακριβώς ο ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών πρέπει να έχει σχέσεις με τα διάφορα μέρη. Οπότε Φυσικά και θα είμαι προσεκτικός για να είμαι σωστός, δίκαιος στις σχέσεις αυτές με όλους τους μετόχους. Είτε πρόκειται για μεγάλη, για μικρή τράπεζα και κυρίως όσον αφορά τη σχέση με τα λόμπις. Πώς θα το κάνω, θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, ώστε να διασφαλίσω διαφάνεια στην επικοινωνία μου μαζί τους και το καλό είναι ότι ακριβώς και τώρα στη δουλειά μου υπάρχει μεγάλη διαφάνεια. Οπότε ενθαρρύνω και τον κόσμο να φροντίσει, να με αναγκάσει ακόμα περισσότερο. Θα φροντίσω να υπάρχει σωστή ισορροπία ε, πάντως, παίρνοντας ε, ό,τι αντιδράσεις και ό,τι σχόλια από τα επιμέρους μέλη. Τώρα, στη συνέχεια, αν σας κατάλαβα καλά, ρωτάτε αν πρόκειται για μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είναι μια μεγάλη και δύσκολα μπορεί να διατηρηθεί μια ενιαία αγορά ε, με την συμμόρφωση στο ΕΜΕΛΕ και έτσι κι αλλιώς θα είμαστε τόσο δυνατοί όσο δυνατός είναι ο πιο χαλαρός και αδύναμος κρίκος της αλυσίδας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια καλά συντονισμένη προσέγγιση. Και όχι μόνο μεταξύ των AML, αλλά μεταξύ όλων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις σωστές πληροφορίες. Τώρα, κατάλαβα καλά την επόμενη ερώτησή σας, έχει να κάνει με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, αν θα είναι σε θέση να φέρει σε πέρα στα καθήκοντά της ή όχι. Από τις συζητήσεις που γίνονται μέχρι τώρα, εμείς ε, θα έχουμε περιορισμένους πόρους, τους ίδιους δηλαδή που έχουμε και τώρα, για περισσότερο έργο. Οπότε το θέμα δεν είναι να είμαστε εμείς ένας κεντρικός παράγοντας στην Ευρώπη. Ο ρόλος μας θα είναι συντονιστικός επιπλέον. Είναι αυτό ιδεώδες. Μεσοπρόθεσμα νομίζω πως ναι, πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε αυτό το στάδιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος με το θέμα, αλλά είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Και σίγουρα είναι ένας ε, δρόμος στον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για να είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Στρεμόσα, ευχαριστώ Πρόεδρε Καλτιέρη. Καλημέρα κύριε Κάμπα και συγχαρητήρια. Γιατί στο Στρασβούργο καταφέρατε σε πέντε λεπτά οι συντονιστές να συμφωνήσουμε κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Άρα μας πείσατε στην ακρόασή σα και ελπίζουμε να κάνετε καλή δουλειά στη συνέχεια. Για τα MPL τώρα θέλω κάτι να ρωτήσω, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κάτι το οποίο για μένα είναι ένα ζήτημα που δεν έχει λυθεί. Έχει μπλοκαριστεί η κατάσταση και στις τράπεζες επειδή υπάρχουν διαφορές ανάμεσα ε, στον κίνδυνο, τον ε, επιμερισμένο κίνδυνο. Και ρωτάω, είμαστε εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένω ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων και να οδηγηθούμε σε μια κρίση σαν και αυτή του 2008. Μία από τις έμονες ιδέες μου είναι ο κύριος Ντράγκη, ας πούμε, το 2017 σε μία από τις κράσεις του, εγώ τον είχα ρωτήσει γι' αυτό και είχε πει ότι η πηγή των μη ξυπηρετούμενων δανείων είναι η μη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ε, καθυστερημένες πληρωμές. Ε, ξέρετε, υπάρχει κάτι για πληρωμές σε 30 μέρες σε διάφορες ε, χώρες αλλά σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης συνήθως οι πληρωμές μπορεί να γίνουν και μετά από 500 μέρες μερικές φορές. Έτσι, διάφορες μεγάλες επιχειρήσεις για χρόνια δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην ανεργία πολλοί άνθρωποι, να κλείνουν πολλές μικρές επιχειρήσεις. Και έτσι, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα είπε ο Ντράγκη, έτσι δεν τα είπα εγώ, δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Στην Ισπανία, στην θητεία αυτή που λύγει τώρα, δεν ε, μπόρεσε να εγκριθεί τελικά καμία ρύθμιση κυρώσεων για τις καθυστερημένες ε, πληρωμές. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με ρωτάτε πόσο πρέπει να ανησυχούμε όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και κατά πόσο οι τράπεζες είναι εξοπλισμένες να αντιμετωπίσουν ε, αυτό το φαινόμενο εφόσον ξαναπροκύψει όπως το 2008. Κοιτάξτε, το 2008 είχαμε μια θεαματικά μεγάλη κρίση. Ήταν μια κρίση σαν και αυτή της δεκαετίας του 30. Ε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρχεται τόσο συχνά ή τέλος πάντων όχι πιο συχνά από ό,τι την είχαμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν βέβαια οι κυκλικές διαδρομές ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ελπίζω να μην βρεθούμε σε συστημική πάλι κρίση όσον αφορά τι τράπεζες ε, σύντομα. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχει η κεφαλοποίηση των τραπεζών, ε, υπάρχει η έλλειψη συγκέντρωσης και το θέμα της συγκέντρωσης των δανείων. Υπάρχουν προγράμματα ε, που έχουν εφαρμόσει χώρες μεταρρυθμίσεων που πιστεύω ότι πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να μην υπάρχει πια τέτοια συγκέντρωση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων σε χώρες, σε τράπεζες, σε κλάδους. Τώρα, εγώ συμμερίζομαι την άποψή σας όσον αφορά την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές και τι συμβαίνει με αυτό σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο υπογραμμίζω όχι μόνο ότι υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές, αλλά ότι υπάρχει και κάποια εξουσία στις αγορές τελικά. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι αγοραστές, οι κυβερνήσεις, γιατί και αυτές ε, ε, πολλές φορές δεν πληρώνουν όπως είπατε, δεν θα πρέπει να επιβάλλουν ε, στις μικρές μεσές επιχειρήσεις και άλλους τις δικές τους επιθυμίες γιατί έτσι πλήττεται και ο ανταγωνισμός. Πηγαίνουμε προς μία κατεύθυνση, να το πω έτσι, ε, που θα υπάρχουν πιο αποτελεσματικές πληρωμές. Δηλαδή θα υπάρχουν ε, μικρότερα χρονικά διαστήματα κατά μέσο όρο μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η πληρωμή. Και ελπίζω να μην αυξηθεί αυτό το χρονικό διάστημα σε περίπτωση κρίσης, γιατί αυτό έγινε σε διάφορες οικονομίες. Αναφερθήκατε στην Ισπανία. Ναι, υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Η πραγματική πρόκληση εδώ είναι το να επιβάλλουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για πληρωμές. Είναι πολύ βασικός ένας τέτοιος κανόνας. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η ελευθερία η ε, συμβατική, δηλαδή ότι αποφασίσουν οι δύο πλευρές. Περί αυτού πρόκειται, ότι δύο συμβαλόμενοι αποφασίζουν με δικιά τους ελευθερία. Άρα είναι δύσκολο να τους επιβάλλουμε χρόνους πληρωμών. Οπότε, αυτή είναι η απάντησή μου. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σουρτασούν. Ευχαριστώ κύριε Κάμπα. Τρεις ερωτήσεις έχω σύντομα. Πρώτον, οι δοκιμές αντοχής, κατά τη γνώμη σας, ε, πιστεύετε ότι είναι καλές αυτές οι δοκιμές, γιατί από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Έπειτα, όταν ε, πολλούνται παράνομα κάποια προϊόντα στις δημοσιονομικές ε, αγορές, για παράδειγμα η Σανταντέρ, εμείς δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι, πρέπει να σας πω, με το πώς διαχειρίστηκε το θέμα ο κύριος Ένερη. Από πλευράς λοιπόν της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών, εσείς μπορείτε να εμποδίσετε τέτοιου είδου πρακτικές. Τρίτον, κύριε Κάμπα, και εμείς βλέπουμε προβλήματα όταν βγαίνετε από μια τράπεζα με αρμοδιότητες ρυθμιστικές και πηγαίνετε κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια για να μας ε, αποδείξετε, για να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εδώ. Και έτσι συγκεκριμένα ρωτάω, εξακολουθείτε να είσαστε υπάλληλο στη Σανταντέρ και δεν θα ήταν προτιμότερο να έχετε εγκαταλείψει αυτές τις αρμοδιότητες πριν να είστε υποψήφιος για διορισμό στη θέση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πρώτον, για τις δοκιμές αντοχής. Νομίζω ότι το έχω κάπως καλύψει, αλλά εγώ δεν θα είμαι τόσο επικριτικός όπως ήσασταν εσείς όσον αφορά την επιτυχία ή όχι των δοκιμών έχουν αυξήσει κατά πολύ την διαφάνεια οι δοκιμές αυτές αντοχής και η αντίληψη που έχουμε για το κατά πόσο είναι δυνατή μια τράπεζα ή όχι. Τώρα βέβαια εξαρτάται πώς βλέπει κανείς το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Στόχος των δοκιμών αντοχής είναι να εντοπίσουν τις τράπεζες οι οποίες κινδυνεύουν να κλείσουν που είναι πιο ευάλωτες από άλλες. Και έχω την αίσθηση ότι αν κάνετε τις δοκιμές αυτές και δείτε μετά κατά πόσο οι τράπεζες που κλείσαν ή όχι, πέρασαν ή όχι από τα, από τις δοκιμές αντοχής, εκεί θα δείτε αν όντως φαινόταν ή όχι το πρόβλημα. Πάντα βέβαια υπάρχει και το περιθώριο σφάλματος. Πάντως και ο προηγούμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών το έχει πει ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που θα κάνει αυτές τις αλλαγές. Στον επόμενο κύκλο πάντως εμείς θέλουμε αν μη τι άλλο να υπάρξει αυτός ο προβληματισμός και η συζήτηση. Δεύτερον, όσον αφορά τις ε, πωλήσει τις ε, παράνομες, δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή, μηδενική ανοχή. Τι σημαίνει βέβαια αυτό και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτή η αρχή. Πρώτα απ' όλα, ποια πληροφορία είναι κατάλληλη. Ε, πώς μπορούμε να προβλέψουμε κατάλληλα, ε, κατά πόσο οι εγγύσει θα είναι ικανοποιητικέ ή όχι. Οι πληροφορίες αυτές, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να έρχονται επειδή υπάρχει διαφάνεια καταρχήν σε ένα μεγάλο βαθμό και δεύτερον από το profiling του πελάτη. Αλλά συνολικά η προστασία των καταναλωτών είναι ένα θέμα το οποίο θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία όσο περνάει ο καιρός ήδη τα τελευταία 5-6 χρόνια. Κάναμε τα περιξηγένση τραπεζών, συνεχίζουμε και πιστεύω ότι η προστασία του καταναλωτή θα βρίσκεται πάντα στο κέντρο ε, των ανησυχιών Τώρα για τη σχέση μου με την τράπεζα Σανταντέρ. Βλέπω ότι αυτό ε, σας ενδιαφέρει, σας απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με ρωτάτε τι θα κάνω. Βεβαίως, ευχαρίστως, θα έρθω ξανά και όποτε μου το ζητήσετε να θα ξανάρθω εδώ για να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις ή ανησυχίες έχετε. Αυτή είναι μια προσφορά εξορισμού. Με ρωτήσατε αν εξακολουθώ να είμαι υπάλληλος Ταντερ. Ναι, ετοιμάζομαι να φύγω. Λέτε, δεν θα τα καλύτερα να μην είμαι πια υπάλληλο. Ίσως για την υποψηφιότητά μου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μπορεί, αλλά από την άλλη μεριά έχω μια σταδιοδρομία, έχω μια ζωή, πρέπει να δουλεύω και έτσι καλλιώς δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα, οπότε να παρετηθώ πρώτα, μετά να υποβάλω την υποψηφιότητά μου για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και μετά να μην προχωρήσει, ε, καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος αυτός θα ήταν δυσανάλογος. Μια, ε, δυο, τρεις εβδομάδες αν είχα παραιτηθεί από την τράπεζα Σανταντέρ ε, πριν έρθω εδώ δηλαδή θα είχε κάνει καμιά διαφορά, πιστεύετε. Η σχέση ή τα οποιαδήποτε ε, συμφέροντα δεν πρόκειται αυτό να άλλαζε μέσα σε δύο-τρεις εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την τόσο ειλικρινή απάντηση, το τελευταίο δύσκολο ερώτημα δηλαδή. Νομίζω μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ακρόαση. Αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση. Πολύ σας ευχαριστούμε. Θα κάνουμε μία διακοπή και θα ψηφίσουμε στις 12.30.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Αγαπητέ Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, σας παρακαλώ να αρχίσουμε κάνοντας μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία, ε, αλλά όπως είπα δοκιμαστική, έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ορισμένοι ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε όλες και όλοι. Βάλτε τις ε, κάρτες σας στην κατάλληλη σχισμή του μηχανήματος. Ευχαριστώ πολύ. Θαυμάσια. Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε με τις ε, αναδιαβουλεύσεις για τις εκβάσεις των, ε, για τα αποτελέσματα των ε, τριμερών διαλόγων και πρώτα για το ΠΕΠΣ e η κυρία Ιντφέλτ, την οποία ε, συγχαίρω για την εργασία της στον τριμερή διάλογο, αρχίζει, είναι ονομαστική η ψηφοφορία αυτή. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν για το θέμα με τα αρχικά PEPS, προσωπικά προϊόντα, ε, προσωπικά συνταξιδοτικά προϊόντα. Σας ευχαριστώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Ψήφι 25 υπέρ 4 κατά και 17 αποχές εγκρίνεται και συγχαίρω την εισηγήτρια. Προχωρώ στην έκθεση, στις δύο εκθέσεις του κυρίου Χέκμαρκ. Συγχαίρω και τον κύριο Χέκμαρκ καθώς και τον Πέτερ Σίμων για την σημαντική αυτή διεκπαιρέωση ενός ε, δύσκολου νομοθετήματος. Νομίζω ότι τα πήγατε πολύ καλά. Αρχίζει η ψηφοφορία, όπως είπα, ονομαστική και αυτή. Πέρα της ψηφοφορίας. 44 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 0 αποχές. Συγχαρητήρια. Δεύτερη ε, ψηφοφορία, BRD, αρχίζει ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. 44 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και καμία αποχή, πράγματι ευρύτατη πλειοψηφία, συγχαρητήρια και πάλι. Θα θέλατε να πείτε κάτι κύριε Χέκμαρκ. Ναι κύριε Πρόεδρε, πρώτα θα ήθελα να πω ότι με έχει συγκινήσει η υποστήριξη και κάπω πιο σοβαρά τώρα. Ευχαριστώ όλους τους και ηγητές. Ήταν δύσκολο το θέμα, ωστόσο οι συζητήσεις ήταν επικοδομητικές και στις τελικές ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μπορέσαμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε με πολύ επικοδομητικό τρόπο. Και εσείς κύριε Πρόεδρε τα πήγατε θαυμάσια. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να ευχαριστήσω όλες και όλους τους σκιώδεις, όσοι είναι παρόντες και όλους τους υπολείπους βεβαίως. Ήταν και η τελευταία έκθεση την οποία ξεπώνησα εδώ ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για μένα αυτό είναι πηγή ιδιαίτερη συγκίνησης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πραγματική ευχαρίστηση η συνεργασία μαζί σας και με όλη τη διαπραγματευτική ομάδα. Τώρα, Πέτερ Σίμον. Δύο εκθέσεις του Πέτερ Σίμον. Πρώτον, ERD5, 5 ψήφος αρχίζει. Πέρας ψήφι 41 υπέρ, 2 κατά, 5 αποχές. Δεύτερη, τώρα CRR2, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας, ψήφι 41 υπέρ, 2 κατά και 5 αποχές μεγάλη και ευρύτατη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Σίμων και σε όλη την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να πείτε κάτι, κύριε Σίμων. Πέτερ Σίμων, ευχαριστώ πολύ προς όλες και όλους τους ε, σκιώδης συγητές. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα, διότι μπορέσαμε να δείξουμε ότι και σε δύσκολα θέματα με συνεργασία μπορούμε να ε, καταλήξουμε σε μια ισχυρή ε, θέση του Κοινοβουλίου και εύχομαι σε όλες και όλους οι οποίοι θα ασχοληθούν με την Βασιλεία 3 στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία να επιτύχουν. Τέθηκε και το θέμα στην προηγούμενη συζήτηση με τον υποψήφιο, το θέμα της αναλογικότητας και αυτό θα επανέλθει στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία με πολύ έντονο τρόπο. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία τα τελευταία χρόνια και βεβαίως Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλε και όλου εκείνου οι οποίοι θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Σα ευχαριστώ Πέτερ και συγχαρητήρια και πάλι ο πρόεδρο ε, Γκουαλτιέρη. Πραγματικά θαυμάσια συνεργασία με θαυμάσιους συναδέλφους και θα ε, έχετε κάθε λόγο να είστε υπερήφανος για την έκβαση της εργασίας σας αυτής. Ακολουθεί τώρα, ακολουθούν μάλλον οι διορισμοί. Πρώτο για το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα... Πρώτα, πρώτα η προφορική τροπολογία. Πρώτα ψηφίζει η προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, με μυστική ψηφοφορία, ο διορισμός του κυρίου Λαβιόλα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ψήφι 37 υπέρ, 8 κατά και 3 αποχές με τον κύριο Λαβιόλα. Προχωρώ στο επόμενο θέμα, γνωμοδότηση για τον διορισμό του κυρίου Λέιν ως μέλους τη Εκτελεστική Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει προφορική τροπολογία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Και τώρα θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία για την έγκριση του διορισμού του κυρίου Λέιν ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μια οκταετία με μονομιστική μυστική ψηφοφορία. Πέρας. Ψήφι 33 υπέρ, 8 κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Λέιν. Τέλος, διορισμός του Προέδρου, του, κύριου, του Προέδρου Τη Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, δηλαδή για την υποψηφιότητα του κ. Κάμπα. Υπάρχει πρώτα προφορική τροπολογία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Και τώρα προχωρούμε στην έγκριση του διορισμού του κ. Κάμπα ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για πενταετή θητεία. Με μυστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. 35 ψήφοι υπέρ, 8 κατά, 5 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κάμπα. Θα ήθελα επίση να σημειώσω, λέει ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Α, ναι, μια στιγμή. Πρώτα η κυρία Μπερές και μετά νομίζω ότι θα πούμε τελικά το ίδιο πράγμα, αλλά η κυρία Μπερές πρώτη. Ευχαριστώ. Οι τρεις ορισμοί αυτοί είναι σημαντικοί. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η διαδικασία που ακολουθήσαμε <clears throat> οδηγεί στο να επιλέξουμε ανθρώπους που θα φέρουν σε πέρας ε, καλά τις αρμοδιότητές τους. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Δυστυχώς, εμείς αποφασίσαμε τους τελευταίους ορισμούς για αυτή τη θητεία μας αλλά το θέμα της ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων. Δηλαδή, πόσες γυναίκες υπάρχουν στους υποψήφιους. Είδατε σήμερα το αποτέλεσμα. Η Ντανιέλ Νουή δεν είναι πια πρόεδρος, αντικαταστάθηκε από έναν άντρα στον ESM. Και το ίδιο ισχύει και με τη Σαμπίν Λόξτεμπεργκ από ό,τι έχω καταλάβει. Και αυτή θα εγκαταλείψει τα καθήκοντά της βάση κανόνων που έχουν να κάνουν με την Κεντρική Τράπεζα, έτσι, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι με μας. Είναι λοιπόν ένα μήνυμα αυτό, Πρόεδρε, το θυμόσαστε ότι είχατε γράψει τον Μάριο Σεντένο ακριβώς για να ε, του εκφράσετε την ανησυχία μας για τις ε, συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώνονται οι κατάλογοι υποψηφιωτήτων. Υπάρχει επιτροπή, υπάρχει το συμβούλιο που μας στέλνουν αυτές τις επιλογές, το shortlist. Καλό θα ήταν και εμείς να επιμείνουμε, γιατί μόνο τότε θα μας ακούσουν. Έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να αλλάξουμε την πραγματικότητα και αυτή δεν θα την αλλάξουμε μόνο μιλώντας για το παρελθόν. Πρόεδρος, Πρόεδρος Γκουαλτιέρη, σας ευχαριστώ Περβάνος. Πράγματι σημειώνουμε και εμείς την αντίφαση ανάμεσα στο γεγονό ότι εγκρίναμε τον διορισμό εξαιρετικών υποψηφίων, αλλά για κάθε συγκεκριμένη ατομική περίπτωση υπάρχουν βεβαίω διαφορετικά ιστορικά. Αφενό ε, υπήρχε μία μοναδική υποψηφιότητα και ούτω καθεξής Γνωρίζουμε το ιστορικό αυτό της κάθε υποψηφιότητα. Δεν μπορούμε να επικρίνουμε συγκεκριμένα τις ατομικές αυτές περιπτώσεις. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι η συνολική εικόνα είναι τέτοια που δείχνει ότι συλλογικά η Ένωση δεν έχει επαρκή ικανότητα να προωθήσει την ισότητα μεταξύ των φύλων. Και αυτό είναι ασφαλώς ένα θέμα πολιτικό, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Και η ισότητα φύλων δεν είναι το μοναδικό θέμα βέβαια. Έχουμε και ένα θέμα διαφορετικών προελεύσεων. Μιλήσαμε πριν και για την ανάγκη της διαβούλευσης, ο κ. Λάγκεν είπε κάτι πολύ σωστά. Έχουμε μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις και την ατυχή περίσταση ότι το Κοινοβούλιο, η κοινοβουλευτική θητεία δηλαδή, λύγει πριν να προλάβει να κάνει τις πιο σημαντικούς διορισμούς. Υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Και βέβαια υπάρχει και ένα πολιτικό πρόβλημα. Θα θέσουμε αυτό το ζήτημα ξεκινώντας από συζήτηση με τους συντονιστές για να βελτιωθεί η ικανότητα του Κοινοβουλίου να δώσει πιο ξεκάθαρες κατευθύνσεις ώστε να ενστερνιστούν όλα τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία μια συνολική δέσμευση για την πρόθεση της ισότητας των φύλων στην εκπροσώπηση στα όλα τα θεσμικά όργανα. Έχετε το λόγο, κύριε Γκίλγκουτ. Ευχαριστώ. Γκίλγκολ, συγγνώμη. Δεχθήκαμε τις τροπολογίες που έγιναν για, τις, για τους διορισμούς για να καταστήσουμε σαφέ ότι είναι ένα θέμα αυτό για μα, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα όμω το έχουμε δείξει κατ' επανάληψη και μετά τον τελευταίο διορισμό, τον κύριο Ντεγκίνιο όπως είπατε και εσεί κύριε Πρόεδρε, είχαμε γράψει επιστολή στον κύριο Σεντένο για να ζητήσουμε αλλαγή στην διαδικασία για το πώς γίνονται οι προτάσεις υποψηφιότητων. Όσο τίποτα δεν επιτεύχθηκε ως τώρα. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε να ψηφίζουμε τον ένα άρενα υποψήφιο μετά τον άλλο, θα θεωρηθούμε από το Συμβούλιο λίγο πολύ ως η χρήσιμη ηλίθη δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα τη εξορρόπησης τη εκπροσώπηση των φύλων. Θα πρέπει να θέσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια και να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποιε αλλαγέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω αντίρρηση κατά ιασδήποτε των υποψηφιωτήτων, αλλά χρειάζεται να γίνει μια συγκεκριμένη προσπάθεια για να επιτευχθεί η εξορρόπηση των φύλων και όχι απλώς να καταγγέλλεται. Φέρμπερ, Ψηφίσαμε. Τροπολογίες κατέθεσαν το Λαϊκό Κόμμα και ε, οι σοσιαλδημοκράτες. Και τώρα ακούω ομιλίες και τοποθετήσεις από ανθρώπους που ναι μεν δέχτηκαν την τροπολογία, αλλά αν έχετε διαβάσει τις προφορικές τροπολογίες, όμως αν δεν έχετε εξορρόπηση των εξυπροσωπήσεων στο εθνικό επίπεδο, θα το έχουμε και στο ευρωπαϊκό. Υπήρχε μια ε, κυρία εκπρόσωπος υποψήφια μάλλον και η πλειοψηφία ωστόσο της Επιτροπής Οικονομικών καταψήφισε την υποψηφιότητά της. Δεν μου αρέσει πλέον αυτό, αυτή η συζήτηση βιτρίνας να λέμε «Α, τι φρίκι, τι φρίκι, αλλά όταν εμφανίζεται μια γυναίκα η υποψήφια δεν υπάρχει απολύτως καμία πλειοψηφία υπέρ της ε, υποψηφιότητάς της. Δεν μου αρέσουν λοιπόν αυτά τα υποκριτικά, υποκριτικές τοποθετήσεις. Σβεν Γκίγκολτ των Πρασίνων λέει ότι εμεί υποστηρίξαμε την υποψηφιότητα αυτή. Καλώ. Όλοι είχατε τη δυνατότητα, δυνατότητα να τοποθετηθείτε. Το σωστό και αυτό που ήθελα να πω είναι από το κείμενο το οποίο εγκρίναμε μετά από πρωτοβουλία του Λαϊκού Κόμματο και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, έχουμε γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου με το κείμενο που αναφέρεται ακριβώ σε αυτό το θέμα. Και αυτό που αποφασίσαμε είναι να μην ανακόψουμε την πορεία των υποψηφιωτήτων που είναι καλέ, διότι υπερψηφίσαμε την, ε, τον διορισμό των υποψηφίων αυτών. Από την άλλη μεριά θέλουμε να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Νομίζω ότι είναι μια ξησορροπημένη στάση του Κοινοβουλίου και πολύ σωστά κάναμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τώρα και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των όσων μόλις ψηφίσαμε. Και όπως είπα, κάθε συγκεκριμένη υποψηφιότητα έχει και ένα ιστορικό. Υπάρχει όμως το συνολικότερο πρόβλημα το οποίο θέτουν οι τροπολογίες τις οποίες εγκρίναμε. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και Συντονισμός Οικονομικών Πολιτικών με εισηγητή τον κύριο Βαντεντεν Κέντελάρε. Συμβαστική Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F σιγματάφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H η υπέρ Α, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε. 168, 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M, όλες αυτές είναι οι συμβαστικές τροπολογίες. Α, δεν είμαι στα καλά μου σήμερα, λέει ο πρόεδρος. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. M συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Q υπερκατάποχες κατά αποχές εγκρίνεται. R υπερκατάποχες εγκρίνεται. Συμβαστική S σίγμα υπερκατάποχες εγκρίνεται. Ψηφοφορία επί του συνόλου του τροποποιηθέντος κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Ψήφι 35 υπέρ, 9 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Βαν Ντένκεν Κεντελάρε. Εδώ ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας. Η επόμενη θα γίνει την Δευτέρα 4 Μαρτίου από τις 3 έως τις 4.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη η συνεδρίαση.